et bienvenue à tous. Καλημέρα. Bonjour. Y des objections ou des sur le du À Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για την μερίσια διάταξη γίνονται, ε, γίνεται δεκτής. Τώρα, τα πρακτικά της 28ης και 29ης ε, Μαΐου. Τα έχετε λάβει. Έχετε κάποιες παρατηρήσεις? Αν ναι, θα πρέπει να τις ανακοινώσετε στη γραμματεία μας πριν το τέλος της συνεδρίασης, αλλιώς θα θεωρηθούν δεκτά τα πρακτικά. Τώρα, η υιοθέτηση των αποφάσεων και συστάσεων των συντονιστών, της συνεδρίασης των συντονιστών της 28ης Μαΐου. Μία παρατήρηση να κάνω εδώ, επί των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά με την ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις τροπολογίες και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα πρέπει να γίνεται η αντιληγή απόψεων, υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στην απόφαση των συντονιστών, η οποία ελήφθη στις 28 Μαΐου, και στα αποτελέσματα της γραπτής διαδικασίας η οποία την ακολούθησε. Για να αποφευθεί κάθε σύγχυση, θα ήθελα το συγκεκριμένο θέμα να τεθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασής μας γενικότερα και για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα στο μέλλον, πιστεύω ότι ως συνήθως τα ευαίσθητα θέματα δεν θα πρέπει να γίνουν ε, αντικείμενο γραπτής διαδικασίας, αλλά συζήτησης ανάμεσα σε συντονιστές. Η χρήση της γραπτής διαδικασίας δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην αμφισβήτηση μιας απόφασης που λήφθηκε ομόφωνα ή με συνένεση έστω από τους συντονιστές. Μία επιπλέον ανακοίνωση τώρα. Μία διευκρίνηση στα πλαίσια των ανακοινώσεων της Προεδρίας. Αφορά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του ΣΑΕΛ. Εγώ προσωπικά πιστεύω και πάντα το πίστευα ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει κανείς τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σαχέλ χωρίς να αναφερθεί στα δραματικά προβλήματα της Δυτικής Σαχάρα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τραγικά και να πω ότι σύμφωνα με το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα του πληθυσμού η αυτοδιάθεση θεωρείται θεμελιώδες δικαίωμα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο να ασχοληθεί κανείς με τα δικαιώματα στο Σαχέλ αν δεν ασχοληθεί με τα θέματα της Δυτικής Σαχάρας. Όλα τα πρακτικά, έγγραφα και κείμενα τα οποία δεν αναφέρονται στη γνωμοδότηση την οποία προανέφερα είναι στρεβλά αποδεδόμενα και γι' αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί αυτό το οποίο είπα σε όλους τους ενδιαφερομένους και γραπτά. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρω αν έχει να μας κάνει κάποια ανακοίνωση, όχι. Υπάρχει ένα επιπλέον θέμα με ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για την ερώτηση της κυρίας Γκρέζ, στην οποία, ε, για την οποία θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας δώσει την απάντησή της. Ο κύριος Τζαμάρκο Σκόπα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσω στην ερώτητό σας. Εμείς δεν αναγνωρίζουμε τη μεταβατική κυβέρνηση στη Γουινέα Μπισάου γιατί δεν είναι καρπός δημοκρατικής διαδικασίας. Είναι δύσκολο λοιπόν να πιέσουμε τις αρχές αυτές έτσι ώστε να προστατεύσουν το Βαρέλα National Park. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ασκήσει περιορισμένη διπλωματική πίεση μέσω της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Εθνών και του ειδικού εκπροσώπου του Ηνωμένων Εθνών ε, για την Γουινέα Μπισάου. Όταν υπάρξει δημοκρατική κυβέρνηση τότε θα φροντίσουμε έτσι ώστε η προστασία των οικοτόπων να συμπεριληφθεί στον πολιτικό διάλογο με τις αρχές. Θα εξετάσουμε εν τω μεταξύ και τον ρόλο τον οποίο μπορεί να παίξει η κοινωνία των πολιτών για το συγκεκριμένο θέμα. Κυρία Γκρέζ, έχετε μια παρατήρηση? Όχι. Καλώς, περνάμε τώρα λοιπόν στο επόμενο θέμα, το θέμα 7, πρόκειται για τις προκλήσεις της ε, διμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας ε, στην προοπτική ενός κράτου μέλους και γι' αυτό με μεγάλη χαρά καλωσορίζω στο εσωτερικό της Επιτροπής μας τον κύριο Πασκάλ Καμφά, αναπληρωτή Υπουργό υπεύθυνο για θέματα ανάπτυξης της Γαλλικής Δημοκρατίας. Αγαπητέ Πασκάλ, σας ευχαριστούμε για το ότι είστε μαζί μας εδώ. Θα μας μιλήσετε για τα θέματα της επικαιρότητα στον τομέα της ανάπτυξης και της βοήθειας. Είστε παλαιός Ευρωβουλευτής, γνωρίζετε πολύ καλά το όργανό μας και θα συμφωνήσετε μαζί του ότι έχει σημασία να υπάρχει σωστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων εταίρων στην εφαρμογή και την σύλληψη των ευρωπαϊκών πολιτικών και συγκεκριμένα της πολιτικής για την ανάπτυξη. Οι σωστές σχέσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη είναι θα έλεγα βασικό ε, στάδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της ίδιας και γι' αυτό ο συντονιστής τη Επιτροπή μα, οι συντονιστέ της Επιτροπής μα πήραν την πρωτοβουλία να προσκαλέσουν στην Επιτροπή μα τους εκπροσώπους των κρατών μελών για να ανταλλάξουν ιδέες πάνω στα θέματα που μας απασχολούν στον χώρο τη ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, είναι το θέμα της χρηματοδότησης της δημόσιας βοήθειας για την ανάπτυξη, είτε από την Ένωση είτε από τα κράτη-μέλη. Λυπούμεθα ε, για τη μείωση της βοήθειας αυτής σε ορισμένα κράτη-μέλη και όχι μόνο σε αυτά που θίγονται από την οικονομική κρίση. Οι εξελίξεις αυτές μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην αναφέρει κανείς προς την κατεύθυνση αυτή την ανάγκη μιας πολυοργανικής ε, ε, συμφωνίας για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης 14-20 και τις επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοια συμφωνία στο μέσο χρηματοδότησης της ανάπτυξης για τη συνεργασία και στη χρηματοδότηση της συνεργασίας με τις χώρες ΑΚΕ. Θα ήθελα λοιπόν τώρα, χωρίς να καλυστερήσω άλλο, ε, τον λόγο στον Υπουργό κύριο Κάμφα για να κάνει την εισαγωγή του. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Εύα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα η πρόσκλησή σας και αν κατάλαβα καλά είμαι ο πρώτος Υπουργός Ανάπτυξης μιας χώρας μέλους που ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκλησή σας και ελπίζω να ακολουθηθώ και από άλλους Υπουργούς τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία πράγματι να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις. Σαν τέος μέλος σε άλλες επιτροπές, στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και στην Οικονομική Επιτροπή, γνωρίζω σε ποιο βαθμό οι συζητήσεις ανάμεσα στους εθνικούς υπευθύνους και τους ευρωβουλευτές έχουν μεγάλη σημασία αν θέλουμε πράγματι να ασκήσουμε τις πολιτικές μας με ιδιαίτερη συνοχή και γι' αυτό η πολιτική για την ανάπτυξη είναι μια πολιτική η οποία μοιράζεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη από τη μία και την Ένωση από την άλλη. Εγώ θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή σημαία είναι και η γαλλική σημαία λίγο και η γαλλική σημαία είναι και αυτή ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής σημαίας και γι' αυτό Προσπαθώ συστηματικά να κάνω ό,τι μπορώ έτσι ώστε η συνοχή ανάμεσα στη δική μου δράση ως ο δημοσίου υπευθύνου μιας χώρας μέλους της Γαλλίας και να είναι συμβατή με την δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γαλλία έχει μια δομή βοήθειας προς τις τρίτες χώρες. Τα δύο τρίτα των δωρεών μας πηγαίνουν προς χώρες προς ε, ε, υποανάπτυξη και περνούν όμως από τα δύο τρίτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι λιγότερο από το 20% του ΦΕΔ χρηματοδοτείται από τους Γάλλους φορολογούμενους. Νομίζω λοιπόν ότι τα δύο αυτά ποσοστά από μόνα τους δείχνουν σε ποιο βαθμό οι εθνικές πολιτικές και οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού. Πριν αναφερθώ τώρα σε αυτήν τη μορφή ολοκλήρωσης ανάμεσα στην εθνική πολιτική και την ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της ανάπτυξης, θα πρέπει να εκφράσω κάποιες σκέψεις για τις αλλαγές οι οποίες έχουν αρχίσει να συμβαίνουν στον κόσμο, τις αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν την πολιτική ανάπτυξη και τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζουμε. Καταρχάς και αντίθετα με το τι συνέβη στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στη δεκαετία του 80, δεν ζούμε σε ένα κόσμο όπου να υπάρχουν από τη μία οι χώρες του ΟΣΑ οι οποίες να κυριαρχούν γεωπολιτικά και οικονομικά Υπάρχει θα έλεγα μια αλλαγή στην δύναμη την οικονομική των χωρών η οποία εξελίσσεται. Από τη μία έχουμε τις χώρες του ΟΣΑ, αλλά έχουμε και τις ε, υποανάδυση χώρες, οι οποίες δεν αναδύονται τόσο πολύ, έχουν μάλλον αναδυθεί θα έλεγα και μας έχουν οικονομικά φτάσει. Η πολιτική λοιπόν την οποία ακολουθούμε ε, διεξάγεται στα πλαίσια αυτής της ανάδυσης ενός τμήματος του κόσμου. Αν και η επανεξισορρόπηση αυτή θέτει ορισμένα προβλήματα και σε επίπεδο εμπορικό και σε επίπεδο κοινωνικό και σε επίπεδο περιβαλλοντικό και άλλα. Πιστεύω λοιπόν ότι η αναπτυξιακή μας πολιτική πρέπει να ειδωθεί με αυτόν τον νέο τρόπο. Αυτός ο νέος τρόπος λοιπόν δείχνει ότι έχουν αρχίσει να αυξάνονται και οι συνέπειες της, των κλιματολογικών αλλαγών. Σε μία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και αναφέρεται και σε άλλες μελέτες παλιότερες, δείχνουν ότι η πρώτη απειλή για την ανάπτυξη σήμερα, η πρώτη απειλή για την θνησιμότητα των παιδιών, για την ασφάλεια προμήθειας τροφίμων, η πρώτη απειλή είναι οι κλιματολογικές αλλαγές. Δεν μπορούμε να βλέπουμε λοιπόν να αντιλαμβανόμεθα την πολιτική μας όπως το κάναμε στη δεκαετία του 70 και του 80. Οι κλιματολογικές αλλαγές σε αυτές τις δύο διαστάσεις είναι καθοριστικές. Και γι' αυτό ακριβώς όταν ανέλαβα τις ευθύνες μου εδώ και ένα περίπου χρόνο στη Γαλλία, ξεκινήσαμε τέσσερις μήνες διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών, με όλους τους εκπροσώπους της κοινωνίας αυτής που ασχολούνται με την ανάπτυξη, έτσι ώστε να προσαρμόσουμε την πολιτική μας στις νέες καταστάσεις. Υπάρχει εδώ ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να, να, αντιμετωπίσουμε, ε, θα έλεγα, κατεξαίρεση. το θέμα του Μαλή. Αναφερθήκατε στο ΣΑΕΛ, πρόεδρε. Δεν αναφερθήκατε ειδικά στο Μαλί, αλλά το Μαλί μας απασχολεί ιδιαίτερα σε καθημερινή βάση. Και έχουμε αναλάβει και μια αναπτυξιακή προσπάθεια η οποία είναι ιδιαίτερα ολοκληρωμένη ανάμεσα στη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ξέρετε η Γαλλία σε αυτή την κρίση αντιπροσωπείται σε τρία επίπεδα. Καταρχάς τη στρατιωτική διάσταση, δεν θα ασχοληθώ με αυτήν, την πολιτική διάσταση, έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα προοδού με τη συμφωνία του Ουαγκαντούγκου πριν από δύο μέρες και τη διεξαγωγή εκλογών στο σύνολο του εδάφους της χώρας και την αναπτυξιακή πτυχή. Τώρα για το στρατιωτικό κομμάτι έχουν γίνει σχόλια δεξιά και αριστερά για το τι κάνουν τα κρατημέλη, για το τι κάνει η Γαλλία, για το τι κάνει η Ένωση ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις. Αλλά στον τομέα της ανάπτυξης υπάρχει μια ιδιαίτερως συντονισμένη δράση. Όταν εργαζόμαστε σωστά πρέπει να το λέμε. Για πρώτη φορά λοιπόν στις 15 Μαΐου οργανώσαμε μια διάσκεψη των δωρητριών χωρών στην οποία ήταν συμπρόεδροι ένα κράτος μέλος, η Γαλλία συγκεκριμένα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πρώτη φορά που σε ένα τέτοιο πλαίσιο, σε μια τέτοια περίπτωση, ένα κράτος μέλος και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθύνουν από κοινού την προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας. Αυτό το κάναμε, το πετύχαμε θα έλεγα, γιατί έτσι συγκεντρώσαμε 3,2 δις ευρώ υποχρεώσεων από πλευράς της διεθνούς κοινότητας για τα επόμενα δύο έτη για την ανάπτυξη του Μαλή, για την επιστροφή των δημοσίων υπηρεσιών και την ανάπτυξη των υποδομών. Θα πρέπει λοιπόν τώρα η διεθνής κοινότητα, η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και σε επίπεδο οικονομικό από πλευράς της διεθνούς κοινότητας και σε επίπεδο διαφάνειας και σωστής χρηστής διακυβέρνησης από πλευράς του Μαλή γιατί αυτές οι οικονομικές υποχρεώσεις έχουν ε, ε, θα έλεγα καθοριστεί στα πλαίσια μια σύμβαση η οποία υπεγράφει από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στις Βρυξέλλες πριν ένα μήνα. Θα ήθελα τώρα μαζί με το Μαλή να αναφερθώ και στα δημοσιονομικά, γιατί μου ζητήσατε να αναφερθώ σε αυτά. Η Γαλλία διατήρησε το επίπεδο το αναπτυξιακό της το ποσοστό για τη βοήθεια το 12 και το 13 είναι το ίδιο, 0,46%. Και η δημοσιονομική προσπάθεια, γιατί ξέρουμε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια δεν είναι από μόνη της νομοθετική, ε, δημοσιονομική, ε, μπορεί λοιπόν να στηριχθεί μέσω ε, της μεταφοράς του 10% των εσόδων του φόρου για τις οικονομικές συναλλαγές που δημιουργήσαμε, που θεσπίσαμε στη Γαλλία το 12. Το διευκρινίζω αυτό γιατί έχει γίνει μια μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση, συνεχίζεται η συζήτηση και πρέπει να πάρετε και εσείς θέση. Στα πλαίσια του προσχεδίου του προϋπολογισμού για το 13 που συζητήθηκε στο τέλος του 12, δώσαμε το 10% των εσόδων που προέρχονται από τον φόρο τον γαλλικό για τις οικονομικές συναλλαγές στην ανάπτυξη και έτσι διευκολύναμε την πρόσβαση στην ιατρική προώνια 2 εκατομμυρίων παιδιών της Αφρικής χάρη στα 30 εκατομμύρια ευρώ που πήραμε από τον φόρο αυτό και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι εμείς οι Γάλλοι που μπορέσαμε να δημιουργήσουμε το μηχανισμό αυτό και να στρέψουμε προς εκεί σε αυτό τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο τα χρήματα τα διαθέσιμα θα πρέπει νομίζω αυτή η αντίληψη να κυκλοφορήσει στο σύνολο της Ένωσης. Γίνεται αυτή τη στιγμή η συζήτηση για τον ευρωπαϊκό ε, τέτοιο φόρο, τον φόρο των 11 χωρών μάλλον. Θα πρέπει να πάρετε μέρος στη συζήτηση αυτή, όχι μόνο έτσι ώστε ένα τμήμα του φόρου αυτού να πάει στην ανάπτυξη, αλλά ο φόρος αυτός θα πρέπει να είναι ο ευρύτερος δυνατός και με ποσοστά να είναι τα υψηλότερα δυνατά έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από μερικούς μήνες που είχε πει ότι χρειάζονται 35 εκατομμύρια ευρώ ή μάλλον πιθανά έσοδα είναι 35 ε, conséquent rapporté par exemple au budget annuel du Fed. 340 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι μια μάχη λοιπόν την οποία έχουμε αρχίσει να δίνουμε και για την οποία η επίσημη θέση της Γαλλίας που υπενθύμησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει ένα τμήμα σημαντικό του φόρου αυτού να στραφεί στην ανάπτυξη. Πέρα από τις προκλήσεις των λεγόμενων καινοτόμων μορφών χρηματοδότησης που δεν περιορίζονται στο φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, υπάρχουν και οι λεγόμενες ιδιωτικές επενδύσεις. Γνωρίζουμε αν και ήμασταν δημοσιονομικά σε θέση να προσφέρουμε περισσότερη συμμετοχή από το δημόσιο δημοσιονομικά, αν ήμασταν σε τέτοια δυνατότητα θα εξακολουθούσε να είναι ανεπαρκής και πρέπει να διασφαλίσουμε ιδιωτικές μορφές χρηματοδότησης. Κάτι τέτοιο δεν είναι μόνο ευκταίο, είναι απαραίτητο. Αλλά θα πρέπει οι επενδύσεις αυτές να σέβονται ορισμένε προϋποθέσεις οι οποίες να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη, γιατί αλλιώς μπορεί να δημιουργήσουν πάρα πολλά προβλήματα όπως στον τομέα των ιδιωτικών επενδύσεων στις πρώτες ύλε, όπου δυστυχώς δεν προσφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη του συνόλου της χώρας αλλά προωθούν τις ε, ε, μη χρηστές πρακτικές. Γι' αυτό ακριβώς και έχουμε αναλάβει την υποχρέωση σε ό,τι έχει σχέση από τη μία με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ε, προϋποθέσεις κατά από τις οποίες γίνονται οι επενδύσεις αυτές οι ιδιωτικές και ό,τι είναι εκτός θα έλεγα των δημόσιων μορφών ε, χρηματοδότησης να σέβονται τους ίδιους κανόνες. Δύο παραδείγματα, δύο προκλήσεις καθοριστικές θα έλεγα. Το πρώτο αφορά τη γεωργία. Προφανώς και χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις στον γεωργικό τομέα. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα μαθήματα της κρίσης που ακολούθησε την έκρηξη των πρώτων υλών των γεωργικών το 2007-2008. Θα πρέπει όμως να σεβόμαστε τους κανόνες του Διευτού ΠΟΕ και ε, τους κανόνες του ΟΗΕ της Υπηρεσίας Αρμόδιας για τα Τρόφιμα. Πήραμε λοιπόν τον προηγούμενο Μάιο την εξής απόφαση. Όλες οι επενδύσεις, οι ιδιωτικές στον τομέα της γεωργίας που θα χρηματοδοτηθούν από την Γαλλική Υπηρεσία Εξωτερικής Ανάπτυξης θα πρέπει να σέβονται τις εθελοντικές βασικές αρχές της υπηρεσίας των θύμων του ΟΗΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και να σέβονται επίσης την διαφάνεια των συναλλαγών. Νομίζω λοιπόν ότι ναι πρέπει να πούμε στις επιπλέον επενδύσεις στον τομέα τον ιδιωτικό, τον γεωργικό από πλευράς ε, ιδιωτών, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε κάποιες καταχρήσεις όπως ε, χρήση των γεών μόνο για εξαγωγές κτλ. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο όχι μόνο σε επίπεδο αρχών αλλά και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμόζουμε έτσι ώστε το δημόσιο χρήμα να μην είναι ο μόνος τρόπος ε, για τις ιδιωτικές επενδύσεις αν δεν γίνονται σεβαστές οι αρχές ε, ε, του Οργανισμού Τροφίμων του ΟΗΕ. Τώρα για τις εξορρυκτικές δραστηριότητες. Χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ευρώπη απέκτησε μια οδηγία αρκετά φιλόδοξη θα έλεγα για τις εξορρυκτικές δραστηριότητες, για τις χρηματοπιστωτικές ε, ροές. Και η διαφάνειά τους στη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και κρατών. Και εμείς υποστηρίζουμε όλες τις πρωτοβουλίες με το στόχο αυτό, όπως ε, άλλωστε δηλώσαμε και στην Τράπεζα Συντήσεων του Συμβουλίου, όπου πιστεύω συμβάλαμε με τη συμπεριφορά μας να αλλάξουν στάση κάποια κράτη που τώρα κάπως πιο διστακτικά. Σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο του G8, σε σχέση με τον Καναδά επίσης, όπου εξασφαλίστηκε δέσμευση αντίστοιχη με αυτή που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν και στο G8 να έχουμε δεσμεύσεις που θα φτάσουν μέχρι την ομάδα των 20, του G20. Και έτσι αυτό που θέλουμε ε, να εξασφαλίσουμε ένα ισότιμο πεδίο, ένα level playing field με το ευρωπαϊκό, το αμερικανικό, μεθαύριο και το καναδικό ε, κείμενο ως βάσης για διαφανή και ευφυή διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από την εξελικτική βιομηχανία. Στον τομέα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής που ξέρω ότι σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, έχουμε λάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες, Δεν επανέλθω εν συντομία και μπορώ να δώσω πιο πολλές λεπτομέρειες αν το επιθυμείτε. Μαζί με την Ορβηγία ήμασταν οι πρώτοι πέρσι που χρηματοδοτήσαμε μια μελέτη σκοπιμότητας της πρωτοβουλίας που ονομάζεται ε, έφορος ή δόε χωρίς σύνορα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πρωτοβουλία, ύστερα από κτηνιάτρους, αγρονόμους και διάφορους άλλους, του εφόρου, του ΣΔΟΕ χωρίς σύνορα, με την καλή έννοια πάντα. Και έτσι, μια πρωτοβουλία που βρίσκεται υπό ε, υιοθέτηση στο Κορεπέρ κατά το τέλος του έτους θα βοηθήσει σε συγκεκριμένους όρους τις χώρες του Νότου να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή. Αυτά είναι διάφορα στοιχεία τα οποία νομίζω δεν έχουν επιβάρυνση για τον προπολογισμό των κρατών. Και επίσης κινούμαστε σε ένα πλαίσιο ευρύτερο, ε, δηλαδή δράσεις πολυαριθμές πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, όπως είπα, για την εξωτερική βιομηχανία, για την ΕΦΕΟ. Ενώ υπάρχουν άλλες πρωτοβουλίες και δράσεις που μπορεί να έχουν δημοσιονομικές, να σημαίνουν δημοσιονομική επιβάρυνση και κυριολεκτόμεθα και για τη σκοπιμότητά τους πολύ πιο σοβαρά. Άρα λοιπόν η πολιτική της ανάπτυξης θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στην ε, κρατική επιχορήγηση για τον ε, προπολογισμό. για την ανάπτυξη δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό δεν αντιστοιχεί πλέον στους ε, σύγχρονους όρους ανάπτυξη αυτού του θέματος και του δημόσιου διαλόγου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να περικοπούν οι Οικονομικέ ενισχύσει. Αλλά θα πρέπει να τι εντάξουμε και να τι εγγράψουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Και εσύ ήμουν εγώ ο πρώτο, ο οποίο ε, έλεγε ότι και το ΦΕΔ και τα άλλα σχετικά εργαλεία, εργαλεία γειτονία δεν θα πρέπει να περικοπούν. Και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονό ότι μπορέσαμε να διατηρήσουμε μακροπρόθεσμα τη δεσμεύση των ευρωπαϊκών κονδυλίων του ευρωπαϊκού προπολογισμού στο θέμα αυτό. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα λοιπόν, αυτονόητο. Αλλά δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο τον προπολογισμό. Γιατί εκεί στελέχουμε πολύ τον ορίζοντά μα. Και αν μου επιτρέπετε, ύστερα από κάποια μηνύματα που ήθελα να απευθύνω, δεν μπορούμε να επανέλθουμε αργότερα στι λεπτομέρειε, στη λειτουργική ε, σχέση μεταξύ κράτου μέλου και Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε να το περάσουμε το θέμα αυτό εν συντομία. Εμεί θέλουμε περισσότερο κοινό προγραμματισμό σήμερα. Την ώρα που έφτανα εγώ στη, που εγω εγώ καθήκοντα, είχαμε 4-5 κράτη με ο πρωτοπόρο δράση. Τώρα είναι περισσότερα αυτά και χαιρόμαστε ιδιαίτερως. Κυρίως δε για τα κράτη στα οποία η ενίσχυση, η ενισχύση που προσφέρει η Γαλλία αλλά και γεωπολιτική παρουσία, η ιστορική παρουσία της είναι πιο σημαντική. Ε, σιγά σιγά ευθυγραμμίζουμε τον προγραμματισμό μας και τον απλουστεύουμε έτσι ώστε να και πιο απλή κατάσταση και για τους εταίρους και ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων ενισχύσεων. Επίσης, αναλαμβάνοντας καθήκοντα επέμεινα ιδιαίτερα ώστε α, και ας είναι το ΦΕΔ εκτός προϋπολογισμού να ε, αφοιερώνεται ένα 20% στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής, γιατί θα ήταν παράδοξο βέβαια να πιέζουμε σε διεθνές επίπεδο για τους περίφημους στόχους Τη βιώσιμη ανάπτυξη το θεματολόγιο για μετά το 2015 δηλαδή, που η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα πριν από μερικέ εβδομάδε με του Υπουργού τη ανάπτυξη, υιοθέτησε μια πρόταση για σύγκληση των δύο αυτών θεματολογιών και από την άλλη όταν κάνουμε τον προγραμματισμό για την περίοδο 2014-2020 συγκεκριμένα για το 2015 και μετά, να μην ενσωματώνουμε μέσα σε αυτή την περίοδο το όραμα αυτό, την αρχιτεκτονική αυτή και να αφήνουμε κατά μέρος την κλιματική αλλαγή. Θα ήταν κάτι το οξύμορο, γι' αυτό και ο Επίτροπος Πίμπαλς δεσμεύτηκε, δεν ξέρω σε συγκεκριμένους όρους αυτό πώς θα εκφραστεί, αλλά δεσμεύτηκε το 20% του ΦΕΔ να αφιερώνεται σε στόχους που βοηθούν στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Εμείς έχουμε και πιο φιλόδοξο ακόμη στόχο για τη γαλλική υπηρεσία για την ανάπτυξη. Έχει έναν συγκεκριμένο στόχο με 50% έργων που παρουσιάζουν αυτό που ονομάζουμε συν ε, αποτέλεσμα συν όφελος, συμπληρωματικό όφελος για το κλίμα, δηλαδή η καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής συγκεκριμένα. Αυτό είναι το 50% των έργων που αναλαμβάνει η δική μας η υπηρεσία ένας μεγάλος στόχος για τη Γαλλία και ξέρετε ότι εμείς θα υποδεχθούμε τη μεγάλη διάσκεψη για το κλίμα το Δεκέμβριο του 2015 μια μεγάλη διάσκεψη η οποία θα μας ε, καλέσει να εξεύρουμε λύσεις και συμφωνίες που δεν είχαν βρεθεί στην Κοπεχάγη. Άρα λοιπόν διάρθρωση, εξισορρόπηση στόχων και αποτελεσμάτων αλλά και κλιματική αλλαγή και έτσι και αναθεωρούμε, αναλογιζόμαστε την πολιτική της ανάπτυξης σε πλαίσιο ακριβώς όπου η κλιματική αλλαγή αποτελεί την πρώτη της βάρος της ε, ανάπτυξης και νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ εύστοχη επιλογή. Πρόκειται για μια από τις κύριες προτεραιότητες των επιλογών και του οράματό μου. Και αν θέλετε πιο πολλές λεπτομέρειες για να κλείσω ε, για το τι έχει γίνει του τελευταίου 13 μήνες στη Γαλλία, έχουμε αφήσει έναν απολογισμό στα αγγλικά εδώ στην είσοδο τη αίθουσα και τα γαλλικά, αγγλικά και γαλλικά λοιπόν, για όσους από εσά ακόμη ίσω ξέρετε γαλλικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πασκάλη, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Και τώρα οι βουλευτές Κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για την ε, ευγενή οργάνωση αυτής της συνάντησης. Μήνες τώρα καλούμε να εξασφαλιστεί η παρουσία των αρμόδιων για θέματα ανάπτυξης υπουργών στα πλαίσια της, στο πλαίσιο της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ Πασκάλ που ήρθες και πρέπει να αποτείνω ο φόρο τιμής ε, για τις προσπάθειές του και για τις ε, πληροφορίες που μας έδωσε. Έχω κάποιες προτάσεις αλλά και κάποιες ερωτήσεις. Λέτε ότι δεν πρέπει να περιοριστεί η συζήτηση στο 0,7% και ότι θα πρέπει να λαδώσουμε κάπως το σύστημα ώστε να δουλεύει πιο αποτελεσματικά. Υπάρχει λοιπόν και το 0,7%, αλλά πρέπει και να αναλογιστούμε ολόκληρο το σύστημα και σε αυτό συμμερίζομαι τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν για τα ζητήματα ή τις δράσεις που δεν έχουν ε, επιβάρυνση για τον προπολογισμό. Δεν θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό. Για, την Ευρωπαϊκή, για τη Γαλλική Υπηρεσία Ανάπτυξης και τη δράση της στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είπατε ότι η υπηρεσία αυτή χρηματοδοτεί μόνο έργα ή προγράμματα με φορείς ε, που ακολουθούν και σέβονται τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΦΕΙΟ. Πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά το πρόβλημα είναι πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την τήρηση της, ε, των αρχών αυτών της ΕΦΕΙΟ από άλλους παράγοντες, άλλους φορείς, πέραν της Γαλλίας ή της ε, Σενεγάλης ή όποιο άλλο, εν πάση περιπτώσει, αναμειγνύεται σε κάποια προγράμματα τέτοια, Την έχουμε πλήρη σεβασμό. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τηρούν τις αρχές αυτές και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν τις τηρούν και καλούνται τώρα να τις στηρίσουν και ιδιαίτερα αναφέρομαι στην Κίνα. Πώς μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε αυτή την αλλαγή παραδείγματος ώστε να ε, ακολουθούν όλε αυτέ τις αρχές. Μια δεύτερη ερώτηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη, το ΦΕΔ. Μας είπες ότι το 20% θα πρέπει να αφιερωθεί στο ίν πολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε και εμεί συζητήσει τα θέματα αυτά, χρόνια τώρα μάλιστα, στην υπηρεσία μα, στην Επιτροπή μας, να δούμε δηλαδή το πώς τα κονδύλια που επενδύονται για τον περιορισμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής για τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να θεωρηθούν ως συμπληρωματικά κονδύλια θα πρέπει να εγγραφούν στον υφιστάμενο ήδη προπολογισμό της ανάπτυξης. Οι περισσότεροι εδώ στην Επιτροπή μας θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά τα κονδύλια. Το είπαμε και στην κυρία Χιντεγκάρτ που ήρθε να μας ε, δει και να ρωτήσει αν εμεί ω Επιτροπή ανάπτυξη μπορούσαμε να δεχθούμε μέγα μέρο του προπολογισμού αυτού αυτής της ανάπτυξης να αφιερωθεί στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αυτά είναι τα ερωτήματα και θέλω να ρωτήσω σε ποιο βαθμό συμφωνείς μαζί μας, Πασκάλ, σε αυτές τις θέσεις. Μια τελευταία παρατήρηση. Περίπου 12 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν τα πάντα για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους με 0,7% συγκεκριμένα. Άλλες χώρες βεβαίως θα έχουν και κάποιες δικαιολογίες ε, ε, όπως η κρίση ή και σοβαρές αιτίε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να έρθουν εδώ και να μας εξηγήσουν γιατί δεν τηρούν το 0,7% και θέλουμε να έρθουν εδώ για να συζητήσουμε ειλικρινά μέχρι πόσο μπορούμε να στύψουμε αυτή τη λεμονόκουπα. Η παρουσία σου εδώ σήμερα έχει τη θέση της αυτήν προσπάθεια να ε, κάνουμε τις χώρες αυτές να αλλάξουν συμπεριφορά. Και μια και σε θεωρούμε σύμμαχο, θέλουμε να μας δώσει συμβουλές για το πώς θα μπορούσαμε να αλλάξουμε αυτή τη συμπεριφορά των κρατών. Ευχαριστώ κύριο Σπέρμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ της Ανάπτυξης της Γαλλικής Δημοκρατίας. Πολύ καλό το ότι ήρθατε και ελπίζω να σας ακολουθήσουν και άλλοι υπουργοί. Το έχουμε περάσει στον ελληνικό από ό,τι κατάλαβα. Μεταξύ μας είμαστε. Είμαστε και πρώην συνάδελφοι, πώς να το πούμε. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε στην Γαλλία, τη Γαλλική Δημοκρατία. Την σεπτή αυτή κυρία. Και θα ήθελα να κάνω τις εξή παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Πέντε το σύνολο, Πασκάλ. Ή μάλλον όχι, να το πιάσω αλλιώς. Έχουμε κάποιοι βουλευτές ε, υποβάλει την πρόταση για την, τον εορτασμένο Ευρωπαϊκό έτους για την ανάπτυξη του 2015. Συζήτηση, διάλογο, αναλογισμό, προτάσεις για την ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την ιδέα αυτή και φαινόταν ότι προχωράει καλά, πλην όμως τώρα φαίνεται πως ορισμένα κρατημέλη εκφράζουν αμφιβολίες για τη σκοπιμότητα της επιλογής αυτής. Η Γαλλία συγκαταλέγεται στα κράτη αυτά. Πώς το κρίνεται σε αυτό, πώς κρίνεται η συμπεριφορά των κρατών αυτών και θα πρέπει να την καταγγείλουμε. Ποια είναι, κύριε πάνω απ' όλα. Βοηθήστε μας λοιπόν. Πρώτο πρώτο αυτό λοιπόν, η κυβέρνηση στη Γαλλία, στο Παρίσι, τι γνώμη έχει και ε, αν δέχεται να συστήσει το 2015 ως έτος για το μέλλον της ανάπτυξης. Επίσης, ναι, μπορεί να υπάρχουν προς τώρα χρήματα, αλλά το 0,3% πότε θα το τηρήσει η Γαλλία. Τρίτον, σύντομη ερώτηση όπως είδες και απλή, σαφής. Η διαφοροποίηση. Η Γαλλία, η Ευρώπη, δεν θέλει πλέον να προσφέρει αναπτυξιακή βοήθεια σε χώρες που παρουσιάζουν πιο μεγάλο ΑΕΠ, Μπορεί εμεί ω Ευρωβουλευτέ να έχουμε αλλάξει κάποια κριτήρια, αλλά εν πάση περιπτώσει χώρε όπω η Ινδία μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνε του. Πλην όμω. Πλην όμω, και εν πάση περιπτώσει θέλω να ρωτήσω αυτή την διαφοροποίηση πώ την κρίνει η Γαλλία. Τέταρτη ερώτηση. Ω εισηγητή για την ε, αναπτυξιακή βοήθεια τη Ένωση, έχω ιδιαίτερα δώσει έμφαση στον αναπτυξιακό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα πρέπει να αξιοποιήσει πολύ περισσότερο το πολιτικό της ειδικό βάρος και τη δυναμική αυτού πολιτικού βάρους, γιατί δεν ε, αντιστοιχεί στο 27% μόνο που βλέπουμε στα χαρτιά, ε, και κυρίως να επιμείνει ας προς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κατανομή ρόλων λοιπόν μεταξύ κρατών μελών και Ευρώπης, πώς σας φαίνεται. Οι κάτω δυστυχώ δυστυχώς περιέκοψαν τον προπολογισμό τους κατά το 1 τέταρτο, δυστυχώς. Ε, επέλεξαν όμως να προσδώσουν στην Ευρώπη αυτό το ρόλο, να είναι δηλαδή η φωνή της δημοκρατίας, των ανθρωπινών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου. Θα ήθελα σε αυτό να προσχωρήσει και η Γαλλία. Τι σκέφτεστε γι' αυτό. Και επίσης τελευταίο με την κυβέρνηση αυτή την καινούρια η Γαλλία τι φρονεί για τα κράτη ΑΚΕ. Πρόκειται για μια έννοια πιστεύω πολύ παροχημένη, μια έννοια ε, που στηρίζεται στην απεικιοκρατική θεώρηση και όχι σε αντικειμενικά κριτήρια φτωχεία ή άλλα. Δεν αποτελεί δηλαδή μια έννοια διεθνών σχέσεων πάνω στην οποία μπορούμε να στηριχθούμε και να αναπτύξουμε υγιείς δεσμούς. Η Γαλλία λοιπόν για την κατάσταση αυτή τι γνώμη έχει. Μαζί με τα κράτη ΑΚΕ που γνωρίζουν όλα άριστα ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και 60 χρόνια μετά μπορεί να μην είναι πια ε, απικίες ορισμένα από αυτά, αλλά ίσως για κάποιους άλλους λόγους, ο οποίος θέλω να επισέλθω, να βρίσκονται σε μια δυσμένη στριχθέση. Εν τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέζ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ έχω ένα μικρό οπλοστάσιο ερωτήσεων. προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ευχαριστώ τον Πασκάλ Καλφά για την δέσμευση και την αφοσίωσή του. Δράτω με τις ευκαιρίες, για να τονίσω πόσο σημαντικά είναι αυτά που μας παρουσίασες, ε, κυρίως στην προσέγγιση της Γαλλίας ως προς την αναπτυξιακή πολιτική που δεν περιορίζεται σε δημοσιονομικά ζητήματα και στην οικονομική αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, η παρουσία σου είναι ειλικρινής και αποσταθεροποιείως. Εκ τούτου θα ήθελα κι εγώ σε σχέση με τους αδέλφους να προσθέσω κάποια πράγματα. Γνωρίζουμε ότι αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να είναι βιώσιμη, για να είναι βιώσιμη και η βοήθεια και γι' αυτό πρέπει να επικρατήσει σύνοχη σε αυτό το τομέα και αυτή τη γραμμή ακολουθούμε από την αρχή της τωρινής θητείας στο Κοινοβούλιο. Ρωτώ το εξή. Ένας Γάλλος υπουργό. ποια δράση μπορεί να αναλάβει το ώστε να αναδειχθεί σε προτεραιότητα αυτή η ανάγκη συνέπειας ως προς την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, βιοπειρατεία. Είχα παρουσιάσει μια έκθεση πρωτοβουλία στο Κοινοβούλιο που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια και καταργώντας έτσι ένα ταμπού. Σήμερα όμως ε, θα πρέπει να κυρωθεί και να υλοποιηθεί το πρωτόκολλο του Ναγκόγια. Δεν εξεπλάγινε δυστυχώς όταν διαπίστωσα την ε, έλλειψη σταθερότητας ως προς την πολιτική της Επιτροπής για τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες και ρωτώ συγκεκριμένα η Γαλλία πώς θα τοποθετηθεί σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομοθετικού χαρακτήρα προτίθεται να δεχθεί αυτή την πρόταση διότι ε, ε, είναι δυσμενής ως προς τη θέση των αναπτυσσομένων χωρών το τονίζω. Τρίτον, Μπέλο Μόντε. Πρόκειται ε, το, για το τρίτο σε τάξη ως προς ε, το μέγεθος του, το φράγμα μετά... Ε, και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για μετακίνηση των δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων αν τελικά οικοδομηθεί αυτό το φράγμα. Πρόκειται για άλλη μία ε, ενεργειακή επιλογή και εδώ και χρόνια όσοι παρακολουθούν το ζήτημα γνωρίζουν ότι οι ευρωπαϊκές και γαλλικές επιχειρήσεις όπου οι Alstom συμμετέχουν στο πρόγραμμα διότι θα έπρεπε να έχουν αποσυρθεί εδώ και καιρό διότι έχουν ε, σημειωθεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βάσει του ποινικού δικαίου. Είχα ειδοποιήσει την κυρία Άστον και με την Εύα Ζολή είχαμε αναφερθεί σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε πάρει πάρα πολύ φλού απαντήσεις ε, προς το παρόν ε, για το ζήτημα αυτό. Ποιο περιθώριο ελιγμών υπάρχει για να παρακινήσουμε τις γαλλικές εταιρείες να αποσυρθούν από αυτό το πρόγραμμα που συνιστά οικονομική και περιβαλλοντική αλλά και κοινωνική καταστροφή για τους γηγενείς πληθυσμούς ε, θυσιάζοντας τον πληθυσμό στο βωμό του της ιδιωτικής οικονομίας, με ποιο τρόπο μπορούμε να έχουμε μια ουσιαστική κοινωνική εταιρική ευθύνη των ευρωπαϊκών και συγκεκριμένα των γαλλικών επιχειρήσεων. Και τέλος, τελευταίο ερώτημα, για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς θα ήθελα να ε, σε ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερους για τα όσα έχεις κάνει στον τομέα αυτό σε συνδυασμό με ε, την ε, Γαλλική Υπηρεσία για την Ανάπτυξη που αποφάσισε πλέον να μην ε, χρηματοδοτεί πλέον έρευνα, αγορά, σπορά και αναπαραγωγή τέτοιων οργανισμών στην Αφρική. Πάρα πολύ καλό όμως υπάρχουν σοβαρότατες αντιφάσεις διότι ήρθε ο Bill Gates πρόσφατα ε, ε, επενώντας ε, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, στον αγώνα κατά της φτώχειας. Διότι συνειδητοποιείται ότι οι γεωργοί θέλουν να ελέγχουν τους σπόρους που χρησιμοποιούν και οι εταιρείε του Bill Gates έχουν εισάγει ήδη τέτοιους οργανισμούς στην Αφρική. Ποια η θέση του Γαλλικού Οργανισμού για την Ανάπτυξη και ποια η θέση θέση των ομολόγων σας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Βανσάν Γκριμό από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Πασκάλ Καλφά για την παρουσίαση που μα έκανε. Θα ήθελα και εγώ να κάνω τρεις σύντομε παρατηρήσεις, δεν θα θέσω επιπρόσθετα ερωτήματα προς το παρόν τουλάχιστον. Πρώτη παρατήρηση Υπάρχει σύγκληση απόψεων ανάμεσα στη γαλλική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τη συνέπεια που χρειαζόμαστε και τη συνοχή στην αναπτυξιακή πολιτική. Χάρη στο Κοινοβούλιο και τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει σημειωθεί πρόοδος, όμως ε, μεγάλο έργο υπολείπεται σε διεθνές επίπεδο. Θα πρέπει να επεξεργαστούν περαιτέρω τα ζητήματα. Επίσης, ε, σε κάποια κράτη-μέλη πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες και τις δράσεις που ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να επικρατεί αποκτήσει συνέπειος προ την εθνική αναπτυξιακή πολιτική ε, των κρατών μελών. Ε, δεύτερη παρατήρηση, σε σχέση με την ε, χρηματοδότηση. Δικαίως ε, μας εξηγήσατε ότι η αναπτυξιακή πολιτική δεν μπορεί να περιοριστεί στα κονδύλια που κινητοποιούνται. Παρόλα αυτά έχουν αναλυφθεί δεσμεύσεις και βλέπουμε να σκιαγραφείται μια νέα, ένας νέος προσανατολισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να φτάσουμε το 0,7% για το σύνολο των δωρητών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αυξήσει τα κονδύλια της. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε και έχουμε εξάλλου και την καταληκτική ημερομηνία του 2015 που ασκεί χρονική πίεση. Τρίτο θέμα. Ε, είπατε ότι είναι σημαντικό να γίνει συλλογικά η προσπάθεια. Πρόκειται για πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κράτη-μέλη. Μιλάμε για πάνω από 40 χώρες ε, και πάνω από τις μισέ ε, θα συντονίσουν τη δράση του στον τομέα της αναπτυξιακής ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και επιχαίρουμε. Επίσης, συλλογική προσπάθεια μας είπατε ναι, αλλά όχι μόνο στην Ένωση, αλλά και στους διεθνείς οργανισμούς. Ε, ε, ο ΙΕ, ο ΩΣΑ, ε, το σύνολο των κρατών μελών θα πρέπει να παίξουν μαζί σαν ομάδα στο πλάι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να προβληθεί η δράση μας σε διεθνή φόρα, όπου είναι και μεγαλύτερα τα διακύβευματα. Σα ευχαριστούμε, λέει η πρόεδρο. Αγαπητέ Πασκάλ, θα σου δώσω το λόγο για να απαντήσεις ε, στις ερωτήσεις και να κάνεις καταληκτικές σου παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για όλα τα ερωτήματα που μου θέσατε ε, πολύ εύστοχα ε, τα περισσότερα και κάποια προκλητικά λίγα όμως και με την καλή έννοια θα επανέλθω στα δημοσιονομικά ζητήματα διότι επικράτησε αυτό το ερώτημα σε διάφορες παρεμβάσεις συναδέλφων Έχουμε περιέλθει σε μια κατάσταση όπου για να επιτύχουμε το 0,7% μας χρειάζονται επιπρόσθετα 4 δις. Σήμερα, δεδομένων των δημοσιονομικών ε, περιορισμών που υπερψήφισε και το Κοινοβούλιο, όπως και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, δεν ε, έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε στο τραπέζι άλλα τέσσερα δις, ε, ενώ ταυτόχρονα έχουμε τα προβλήματα αγοράς εργασίας, συντάξεων και το καθεξής. Ε, υπερβαίνοντας το χάσμα, ε, έχω την εντύπωση ότι σήμερα υπάρχει πλήρης έλλειψη κατανόησης στην γαλλική κοινωνία αν πούμε ότι περικόπ οι κοινωνικές δαπάνες, αλλά διοχετεύουμε επιπρόσθετα τέσσερα δίσες στην αναπτυξιακή πολιτική. Δηλαδή, εγώ ο ίδιος ως υφυπουργό δεν μπορώ να με φανταστώ ε, να ανακοινώνω κάτι τέτοιο. Ε, και πέρα από τα λογιστικά ζητήματα, τίθεται λοιπόν αυτό το ζήτημα συνέπεια. Ε, εάν τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέρα από τις εθνικές δεσμεύσεις, ανέλαβε, αναλάμβανε ε, να ακολουθήσει τα κριτήρια του Μάστριχτ, αντί να μιλάει μόνο για τα εθνικά κονδύλια, θα μπορούσαμε εύκολα να φτάσουμε το 0,7%. Δηλαδή, ε, φάσκει και αντιφάσκει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη θέση που υιοθετεί. Το, οι Βρετανοί αυτό κάνουν και ξέρετε δεν μας συμβαίνει συχνά να χαιρετίζουμε αυτά που κάνουν οι Βρετανοί ομολογοί μας. Ε, πέρα από αυτά που συνέβησαν ε, στην ομάδα G8, που είναι όντως ε, μια πραγματική πρόοδος, ε, ως προς τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις θα πρέπει να τονίσουμε ότι έχουν γίνει προσπάθειες και θα πρέπει να μας προβληματίσει αυτό το ζήτημα. Το πολιτικό κόστος της κυβέρνησης για να τηρήσει τη δέσμευσή της, ε, διότι ένα τμήμα της πλειοψηφίας το προσάπτει στην κυβέρνηση. Η Βρετανική κοινωνία παρόλα αυτά φαίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι η πιο ανοιχτή σε σχέση με αυτή την προβληματική. Εκείνη υπάρχουν ισχυρότερες μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, υπάρχει ε, διακομματική συνένεση, το πολιτικό πολιτικό και το κοινωνικό οικοσύστημα είναι πολύ προηγμένο. Φανταστείτε σε άλλες χώρες που δεν ισχύουν αυτά, είναι σχεδόν ανέφικτο να φτάσουμε το 0,7%. Εντάξει, μπορώ να σας ε, δείξω με λογιστικό τρόπο πώς ακριβώς θα φτάσουμε το 0,7%. Το θέμα είναι πώς θα δημιουργηθούν όμως οι συνθήκες στην κοινωνία, πώς θα το δεχτεί η κοινωνία αυτό και κυρίως ε, πώς θα ε, δημιουργηθούν ε, οι κατάλληλες δημοσιονομικές προϋποθέσεις γιατί όλα αυτά εγγράφονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και ασχολούμαι τώρα μόνο με το παράδειγμα της Γαλλίας και δεν θα αναφερθώ σε άλλες χώρες όπου έγιναν μαζικές περικοπές στις κρατικές δαπάνες. Ε, εξού και η σημασία των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων ε, στον ε, δημόσιο διάλογο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και τη διάθεσή του εν μέρει για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακής πολιτικής, διότι αυτά τα ποσά είναι σχετικά υψηλά και αμήνυμα μόνο θα καλύψουν απώλειες που θα σημειωθούν σε άλλα κονδύλια. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ιερά κάποια κονδύλια, αλλά για την αναπτυξιακή πολιτική μας λέει ότι αν τα κράτη-μέλη αυξήσουν τη συμβολή τους ε, στο ΦΕΔ, θα αντισταθμιστεί αυτό σε άλλα κεφάλαια του προϋπολογισμού. Εντάξει, αλλά αυτό δεν αρκεί. Ε, ως την συνέπεια πρέπει να χαρακτηρίζει τη δράση μας. Ε, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι σε λίγες μέρες θα έχουμε την ε, πρώτη διυπουργική σύσκεψη για την ανάπτυξη τα τελευταία πέντε χρόνια. Ε, εδώ και μία πενταετία η γαλλική κυβέρνηση δεν είχε συγκαλέσει ούτε μία φορά τους συναρμοδίους υπουργούς γεωργίας, οικονομίας, οικονομικών, ε, αλληλείας, περιβάλλοντος για να εξασφαλίσει οχή της δράσης μας. Ε, στον τομέα αυτό. Ε, καταλαβαίνετε πόσο μακρά ήταν και η διπουργική διαδικασία για να οργανωθεί μια τέτοια σύσκεψη. Θα λάβει λοιπόν χώρα. Πέραν αυτού, το φθινόπωρο θα ψηφιστεί ο πρώτο γαλλικό νόμο για την ανάπτυξη. Ολόκληρη την ε, ιστορία τη τωρινή γαλλική δημοκρατία. Επιθυμούμε Α, και να θυμίσω εδώ ότι το έχουν ζητήσει ε, βουλευτές ε, συγκεκριμένα να έχουμε έναν εισηγητή για το ζήτημα της ε, συνέπειας της πολιτικής μας. Όπως αυτό συμβαίνει ήδη στο Βέλγιο. Θα διοριστεί μία, ένα κλιμάκιο βουλευτών που κάθε εβδομάδα θα πραγματεύεται ένα ζήτημα ε, κάποιας πολιτικής, γεωργικής, οικονομικής κτλ. και θα παρακολουθεί την συνέπεια της δράσης ε, των συναρμοδίων ε, Υπουργείων. Ε, και εδώ επαναρχόμαστε στο θέμα της χρηματοδότησης καταπολέμησης ε, των, των κλιματικών αλλαγών. Ε, εξυπακούεται ότι οι χώρες που δικαιούχοι της βοήθειας το αντιλαμβάνονται αυτό ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες οι δύο μορφές χρηματοδότησης. Όμως υπάρχουν και αντιφάσεις. Θα βάζουμε ένα ευρώ για να ε, καταστραφεί το κλίμα διότι αναπτύσσεται η χώρα και μετά θα βάλουμε άλλο ένα ευρώ για να διορθώσουμε τη ζημιά του πρώτου ευρώ. Ε, πρέπει λοιπόν ε, να αναρωτηθούμε πέρα από την προσθετικότητα, την έλλειψη προσθετικότητα των χρηματοδοτήσεων για το ίδιο το περιεχόμενο. Γιατί είναι μεγάλο το διακύβημα οι κλιματικέ αλλαγέ, και πρέπει οπωσδήποτε να συνδυαστεί η πολιτική μας αυτό με την αναπτυξιακή μα πολιτική. Η ενσωμάτωση λοιπόν της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών στην αναπτυξιακή πολιτική θεωρείται από την Παγκόσμια Τράπεζα ως η πρώτη απειλή κατά της αναπτυξιακής πολιτικής. Εγώ αντίθετα πιστεύω ότι το αναπτυξιακό μας θεματολόγιο θα πρέπει να αναδείξει προτεραιότητα το ζήτημα των κλιματικών αλλαγών. Ε, για να είναι βιώσιμη η πολιτική και ένας βασικός άξονας αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει να είναι ακριβώς η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Και βάσει απόφαση του περασμένου Οκτωβρίου για τα ενεργειακά ζητήματα, διότι ε, έξι δι τα επόμενα τρία χρόνια θα διοχετευθούν στον ενεργειακό τομέα. Τα τρία πρώτα είναι για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, συνέχεια ενεργειακή αποδοτικότητα και δεν θα χρηματοδοτούμε πλέον ε, α, α, ε, άθρακα, τις εκπομπές αν ε, δεν υπάρχει δυνατότητα φιλτραρίσματος και αποθήκευσης. Ε, θα διοχετεύσουμε λοιπόν τις επενδύσεις εκεί όπου χρειάζονται περισσότερες ε, υποδομές. Ούτως ή άλλως δεν θα έχουμε τα απαιτούμενα οικονομικά εργαλεία ακόμη και αν κάνουμε τις καλύτερες και τις πιο βαρύγδες πολιτικές δηλώσεις δεν μπορούμε να βάζουμε ένα ευρώ για να καταστρέψουμε το κλίμα και μετά να το αντισταθμίσουμε με ένα ευρώ για να το φτιάξουμε. Αυτό θα είναι κάτι το ιδιαίτερα ευφυές και για τα δημοσιονομικά της κάθε χώρας. Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις νέες πολιτικές μας με την υπηρεσία ανάπτυξης στη Γαλλική και πόσο μπορούν να ενσωματωθούν και στις πρακτικές των άλλων χωρών, θέματα όπως η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων ή τα θέματα που θέτει ο Διεθνής Οργάνος Τροφίμων του πριν πούμε στους άλλους πρέπει να κάνετε αυτό, πρέπει να το κάνουμε πρώτοι και μόνοι μας. Αυτό κάναμε λοιπόν στον τομέα της ενέργειας, της γεωργίας, προσπαθούμε να το κάνουμε στον τομέα της βιοπικιλότητας, του δάσους. Αυτή τη στιγμή στο κάνουμε αυτό, περνάμε στην ενδιάμεση, στη δεύτερη φάση, ζητώντας και από τους άλλους να το κάνουν, γιατί η πραγματικότητα των σχεδίων χρηματοδότησης και της Γαλλικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης, αλλά και άλλων υπηρεσιών, όπως της Γερμανικής, της Λουξεμβουργιανής ή άλλων... ...είναι η μέθοδος πολύ συχνά της συγχρηματοδότησης. η γαλλική υπηρεσία θα θέσει κάποιους κανόνες, αλλά αν οι άλλες οι υπηρεσίες δεν έχουν τους ίδιους κανόνες, σημαίνει ότι ή οι μεν ή δε θα παραβιάσουν τους κανόνες τους. Γι' αυτό ακριβώς και ξεκινήσαμε μια, θα έλεγα, διαδικασία προώθησης αυτών των πρακτικών έτσι ώστε οι κανόνες αυτοί να εφαρμόζονται από κοινού. Κάθε χώρα από μόνη της θα αποφασίσει αν θα δώσει τη μάχη αυτή. Στα γενετικά τροποποιημένα δεν υπάρχει καμία συνένεση. Αναφερθήκατε στο Ίδρυμα Gates και υπάρχουν και άλλοι εταίροι με άλλες απόψεις. Είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο δεν πρόκειται να βρούμε μία συνένεση τους επόμενους μήνες αλλά στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Οι βασικές υπηρεσίες ανάπτυξης συνεργάζονται με την Παγκόσμια Τράπεζα πάνω στον τομέα της ενίσχυσης των κοινωνικών κριτηρίων λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αυτό είναι συμβατό με τις αξίες μας αλλά και με τα συμφέροντά μας. Εμείς θέλουμε η παγκοσμιοποίηση να στοχεύει προς τα όταν χρηματοδοτούμε ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό δεν θα πρέπει να υπάρχουν πρακτικές ασύμβατες με αυτά τα οποία πρεσβεύουμε. Δεν θα πρέπει να πέφτουμε σε τέτοιες αντιφάσεις και γι' αυτό αν το κάνουμε θα μας κατηγορήσει και ο φορολογούμενος, ο Ευρωπαίος. Είναι όμως συμβατό και με τα συμφέροντά μας, γιατί αν πράγματι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οφείλουν να σεβαστούν κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνουν ανταγωνιστικότητα στα εδάφη στα οποία λειτουργούν. Αν εμεί λοιπόν θέτουμε κανόνες στις δημόσιες προμήθειες, διαγωνισμού λέγοντας ότι για να μπορέσετε να πάρετε μέρος ε, στις διαδικασίε ε, του ε, Ιαπωνικού Ντάικα ή της Παγκόσμιας Τράπεζας, θα πρέπει να σέβεστε ορισμένου κανόνε, περιβαλλοντικού και κοινωνικού. Αν είμαστε οι μόνοι που το κάνουμε αυτό, είναι κακό. Αν πείσουμε και τους άλλους αυτό θα μας ευνοήσει. Είναι συμβατό και με τις αξίες μας λοιπόν και με τα συμφέροντά μας. Θα ήταν ακόμα καλύτερο οι επιχειρήσεις οι οποίες ε, δεν παίζουν το παιχνίδι με τους κανόνες αυτού σήμερα να το κάνουν αύριο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό καθορίζει και τη δική μου δράση. Η βασική ιδέα είναι ότι από τον επόμενο Οκτώβριο δεν θα υπάρχουν προκηρύξεις για προμήθειες της Γαλλικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης που να μην περιλαμβάνουν ρήτρε κοινωνικές και περιβαλλοντικές. Οπότε θα τεθεί άμεσα το θέμα των συγχρηματοδοτήσεων. Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να διαδώσουμε την ιδέα αυτή και ζητώ και από εσά να κάνετε το ίδιο. Για τα θέματα των αναδειωμένων χωρών και οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν. Πράγματι σε αυτή τη φάση αυτό το οποίο κάνουμε και είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν στην Υπουργική Επιτροπή τις επόμενες εβδομάδες να επανεξετάσουμε την στρατηγική μας τη γεωγραφική. Δηλαδή, δεν ξέρω βέβαια ποιο θα είναι το αποτέλεσμα εξορισμού αυτής της διαδικασίας. Υπακούμε σε μία αρχή σήμερα, σύμφωνα με την οποία δεν θα πρέπει να υπάρξει κόστος ανακράτος για ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας που γίνεται σε μια αναδιόμενη χώρα όπως την Κίνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέσαμε για πρώτη φορά το 2010 και δεν αμφισβητείται. Κάθε δάνειο το οποίο δίδεται προς την Κίνα δεν έχει κόστος, δεν έχει επιδότηση από πλευράς του κράτους μέλους. Η Κίνα εφόσον θέλει να χρηματοδοτήσει ένα ε, πρόγραμμα μέσω των αναπτυξιακών ταμείων ε, μπορεί να το κάνει αυτό μέσω της αυτοχρηματοδότησής της από τις ε, αγορές σε μακροπρόθεσμο επίπεδο ή σε πιο βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Και μπορεί να συνοδεύει το δάνειο αυτό με την εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία μιας αναπτυξιακής υπηρεσίας, σαν παράδειγμα για την αηφορία των δημοσίων μεταφορών. Περνάμε λοιπόν ένα πακέτο εδώ και διαχείρισης των προγραμμάτων αλλά και οικονομικών και κοινωνικών αρχών. Είναι κάτι που δεν έχει καμία σχέση με τις επιδοτήσεις που ξέραμε στο παρελθόν. Διαφοροποιούμε λοιπόν την αντιμετώπιση των αναδειωμένων χωρών ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξής τους. Αυτό το οποίο είπατε ε, για την Ολλανδία το εφαρμόζουμε ε, στην Κίνα και σκεφτόμαστε να το εφαρμόσουμε τα επόμενα χρόνια και στην περίπτωση της Βραζιλίας ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξής της. Μιλώντας για την Βραζιλία, δεν θα απαντήσω βέβαια στην ερώτηση της κυρίας Γκρέζ, αλλά να πω ότι δεν υπάρχει δημόσιο κόστος, δεν υπάρχει τρόπος χρηματοδότησης ε, για τη συγκεκριμένη χώρα, αλλά δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε σε μια γαλλική επιχείρηση όταν της το ζητά μια ξένη κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια οικονομική συναλλαγή. Αυτό το οποίο αντίθετα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να εργαστούμε πάνω στα θέματα της νομικής ευθύνης των θυγατρικών επιχειρήσεων σε σχέση με τη μητρική. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει έρθει στην επικαιρότητα μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν στον Παγκλαντές. Πρόκειται ένα θέμα πάνω στο οποίο δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει μόνος του σαν χώρα, Γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω και εσείς σαν Επιτροπή Ανάπτυξης να ασχοληθείτε με αυτό. Σήμερα μια θηγατρική, μια ευρωπαϊκή επιχείρηση, η οποία θα διαπράξει συγκεκριμένες ενέργειες που θα έχουν συνέπειες αρνητικές και για τα πρόσωπα, τα φυσικά και για το περιβάλλον, δεν μπορεί να κατηγορηθεί η μητρική εταιρεία για τις πράξεις της θηγατρικής κάτι το οποίο δημιουργεί μια συμμετρία ευθύνη ανάμεσα σε μια οικονομική παγκοσμιοποίηση από τη μία, η οποία ολοκληρώνεται και σε μια νομική παγκοσμιοποίηση η οποία δεν υπάρχει από την άλλη. Βλέποντας τι έγινε στη Γαλλία με την ομολογία της Έρικα μετά το ναυάγιο της Total, της, του πλοίου της εταιρείας Total, η εταιρεία ήταν ε, για πρώτη φορά κηρύχθηκε υπεύθυνη για ενέργειες τις οποίες δεν είχε διαπράξει. Αλλά αυτό έγινε ακριβώς λόγω της δυνατότητας που είχε να ελέγχει τους υπόλοιπους οικονομικούς εταίρους της αλυσίδας. Λοιπόν, αυτό το οποίο λοιπόν τέθηκε και συζητήθηκε στα πλαίσια της γαλλικής περίπτωσης θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εφαρμόσουμε μόνοι μας γιατί θα δημιουργήσει ανταγωνισμούς. Δεν θα πω ονόματα ανάμεσα σε δύο επιχειρήσεις, μία γαλλική και μία μη γαλλική. Από τη μία υπάρχει το, το νόημα, η έννοια της νομικής ευθύνης και από την άλλη δεν υπάρχει. Θα πρέπει όμως να προχωρήσουμε ο καθένας όσο μπορεί περισσότερο σε εθνικό επίπεδο και αυτό που θα ήταν σωστό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί επιτέλους με το θέμα και η Επιτροπή σας μπορεί να είναι ένας από τους χώρους στους οποίους μια τέτοια συζήτηση μπορεί να γεννηθεί, να προχωρήσει και να πείσει. Για την βιοπειρατεία. Θα σας δώσω μία γραπτή απάντηση. Για το έτος της ανάπτυξης. Η Γαλλία επίσημα υποστηρίζει την ιδέα αυτή. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ατζέντα μετά το 2014 θα είναι ουσιαστικά η ατζέντα μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2014. Και δεν ξέρουμε ακόμα αν η αποφασιστική στιγμή για την τελική συμφωνία θα είναι οι τρεις τελευταίοι μήνες του 2014 ή ε, τρεις πρώτοι του 2015. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να καταστήσουμε το 15 έτος ανάπτυξης. Ακόμα και αν το 2014 θα παίξει πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο. Υποστηρίζουμε λοιπόν την πρωτοβολία αυτή. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη διαδικασία του να ονοματίσω κάποιους και να κατηγορήσω, αλλά δεν ξέρω να σας πω ποιες είναι οι χώρες που μπλοκάρουν τις διαδικασίες στο Συμβούλιο. Για τα ΑΚΕ τώρα. Το θέμα τίθεται για μετά το 2020. Έχουμε κάποιο χρόνο στη διάθεσή μας. Αναφέρεστε σε αυτό το οποίο ονόμασα γεωγραφική στρατηγική. Έχουμε μια ζώνη κατά προτεραιότητα χωρών, η οποία αντικειμενικά θα έλεγα έλκει την καταγωγή στην απεικιοκρατική μας ιστορία. Το ίδιο κάνουν και με την κοινοπολιτεία οι Βρετανοί. Εμείς τώρα λοιπόν ανοίγουμε, γυρνάμε μια νέα σελίδα. Λέμε ότι δεν υπάρχει ιεράρχηση που να οφείλεται ούτε στην ιστορία ή σε κάτι άλλο, αλλά σε αντικειμενικούς παράγοντες και μόνο. Κάτι το οποίο μας επατρέπει να είμαστε παρόντες με το ίδιο επίπεδο σε ένα γαλλόφωνο και σε ένα αγγλόφωνο κράτος της Αφρικής. Απ' την άλλη θα μας πούν ότι για λόγους συνεκτικότητας θα πρέπει να πάτε εκεί που έχετε δίκτυα, που είστε πιο αποτελεσματικοί, εκεί που η θέση σας βαρύνει περισσότερο. Αυτό αντικατοπτρίζει βέβαια θα πούνε άλλοι μια μεταπικιοκρατική εικόνα του κόσμου. Όλα τα επιχειρήματα ακούγονται και από τη μία και από την άλλη, αλλά θα πρέπει να καταλήξουμε εμείς πριν από το τέλος του χρόνου στα πλαίσια του συνολικού νόμου, τον Ιούλιο ίσως, για την ανάπτυξη στη Γαλλία. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρεμβαίνουμε οπουδήποτε είναι απαραίτητο, σε επίπεδο αρχής και μετά τώρα αν εκ των πραγμάτων κάποιες χώρες κατά προτεραιότητα τις αντιμετωπίζουμε λόγω της κοινότητας της γλωσσικής σαν παράδειγμα, ίσως οι δυνατότητες που έχουμε ας πούμε στη Σενεγάλη θα είναι πάντα μάλλον μεγαλύτερες από τις δυνατότητες που έχουμε σαν Γαλλία στο Μαλάουι για διάφορους λόγους. Όχι για να διονίζουμε την απεικιοκρατική περίοδο αλλά για να είμαστε απλά πραγματιστές. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Πασκάλ για τις εξηγήσεις αυτές θέλω να πω ότι με μεγάλη χαρά βλέπω ότι αγώνες στους οποίους και εμείς είχαμε αφιερώσει τις δυνάμεις μας σε άλλες περιόδους τώρα αναλαμβάνονται από το G8 για τους φορολογικούς παραδείσους παραδείγματι αλλά και ο συσχετισμός μεταξύ μητρικής και θηγατρικής εταιρείας Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε λοιπόν με χαρά ότι η Γαλλία είναι στο πλευρό μας. Διαπιστώνουμε του, τις και τα όρια των ε, προσπαθειών και τις προσπάθειες για να διαφυλάξουμε το, τα παρθένα δάση του Αμαζονίου και τις προσπάθειες για το φράγμα Μπελαμόντε και βέβαια την ε, σωστή λειτουργία της εξωτερική βιομηχανίας, η οποία και καταναλώνει πολλή ενέργεια και ζητάει πολλή ενέργεια, που έχουμε εμείς επισημάνει ως πρώτη το πρόβλημα και που παρακολουθούμε τακτικά. Και βέβαια θα πρέπει και τα διάφορα νομικά ε, ευρήματα και πλάσματα δικαίου που υπάρχουν να καταπολεμηθούν. Αυτό είναι ο μεγάλος μας αγώνας. Για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ Πασκάλ που ήρθες να μοιραστεί κάποιες ιδέες και τις ε, δυσκολίες ως προς τη δέσμευση του 0,7 που είχε αναλυφθεί σε διαφορετικά πλαίσια. Πάντως εμείς επιτήρουμε την ελπίδα ότι αυτή η υπόσχεση θα τηρηθεί. Και ότι ίσως να αποδειχθεί και μεγαλύτερη η συστράτευση από ό,τι περιμένει η γαλλική κυβέρνηση. Ευχαριστώ και πάλι που έκανε τον κόπο να έρθει μέχρι τις Βρυξέλλες. Θα περάσουμε στο σημείο 8 της ημερησίας διάταξης τώρα. Έκθεση της ομάδας υψηλού επίπεδου σχετικά με το αναπτυξιακό πρόγραμμα μετά το 2015. Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, έχετε την καλοσύνη της συζητήσεις σας να τη συνεχίζετε εκτός της αίθουσας. Les gens sont contents de se retrouver. Τόση είναι η χαρά που ξαναβρεθήκατε. Continuez quand même. Θα συνεχίσω παρόλα αυτά. Η ομάδα υψηλού επίπεδου λοιπόν κατέθεσε πρόσφατα την έκθεσή τη. On va peut-être les demander de sortir. D'accord. Σας παρακαλώ να αποχωρήσετε από την αυσό. Ό,τι δημιουργήσετε, έχετε να τη συνεχίσετε έξω. Ευχαριστώ. Ομάδα υψηλού επίπεδου λοιπόν για το πρόγραμμα για την ανάπτυξη, αναπτυξιακό πρόγραμμα με το 2015. Η έκθεση αυτή κατέστη δημόσια πριν από λίγο καιρό, μια έκθεση που περιμέναμε όλοι, για το μελλοντικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Πρόκειται για μια ομάδα υψηλού επίπεδου με δύσκολο έργο, με διαφορετικές προτεραιότητες και δεδομένα που θα πρέπει να σωματωθούν στο νέο παγκόσμιο πλαίσιο Αρκετές ανησυχίες έχουν εκφραστεί γιατί κάποια από τα σημαντικά και ενδιαφέροντα στοιχεία δεν τα καλύπτει η έκθεση. Ιδιαίτερα η Oxfam έχει σημάνει προβλήματα και ως προς την αναφορά του αγώνα κατά των ανισοτήτων στην έκθεση και εκφράζεται επίσης ότι δυστυχώς κάποιοι παράγοντες, ο πολυπαραγωγικός, πολυπαραγωγικές διαστάσεις της φτώχειας, οι διαφορές στα εισοδήματα, άνηση ανάπτυξη του ΑΕΠ και άλλα προβλήματα δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς, αλλά προτείνω να κοιτάξουμε και τα διάφορα σημεία της εκθέσεως. Η κλιματική αλλαγή, Φερρυπίν, είναι μία από τις κύριες αλλαγές και τι είδους συνέπειες μπορεί να έχει ως προς τον αγώνα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής η ενσωμάτωση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της φτώχειας που μπορεί να οδηγήσει μια πραγματική μείωση των συγκρούσεων και της βίας αλλά μπορεί και να περιορίσει την ουσιαστική αναπτυξιακή βοήθεια εφόσον δεν καταγράφοντας αυτήν ή ε, εξοπλισμοί. Και επίσης, τρίτο κεφάλαιο, μια τρίτη, μια παγκόσμια εταιρική σχέση με έμφαση στην ανάπτυξη και τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών που πολύ καιρό τώρα απασχολούν την Επιτροπή μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ έχουμε να κάνουμε ένα ορόσημο σε, μια, σε ένα δημόσιο διάλογο που θα φτάσουμε στο 2015 και έχουμε ίσως το χρόνο να προτείνουμε κάποιες βελτιώσεις, αναδιατυπώσεις πριν από την Γενική Συνέλευση και την έγκριση από αυτήν στα Ηνωμένα Έθνη της εκθέσεως. Έτσι λοιπόν, με χαρά βλέπω εδώ τον κύριο Αντώνιο Βυζιλάντε διευθυντή του γραφείου της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Εθνών και του προγράμματος για την ανάπτυξη, καθώς και των ε, αρμοδίων για την Ευρωπαϊκή Task Force, τον κύριο Ρούντι Ντεμέγερ την κυρία Σαλδάνια και τον κύριο Βάντερς που είναι εδώ. Παρόντες, καλώς ήρθατε και παρακαλώ τον κύριο Vigilante να λάβει το λόγο για τα λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι πολύ απλό το έργο να σας παρουσιάσω το, την έκθεσή μας. Πολύ σύντομα λοιπόν γιατί έχει δυναμηθεί αυτό. Και μπορώ απλώς να υπογραμμίσω κάποιες εταιρότητες και νέα στοιχεία που περιλαμβάνει. Επιτρέψτε μου πάντως να πω ότι οι στόχοι για την περίοδο μετά το 2015, είτε είναι τη χιλιετία, είτε στόχοι της ανάπτυξης όπως ονομαστούν, ε, σημαίνουν και περισσότερη συμμετοχή, συμμετοχική προσέγγιση, διαβουλεύσεις και νέες τεχνολογίες. Έχουμε παραδείγματι μια ε, επικοινωνία μέσω του διαδικτύου επιγραμμική για να συλλέξουμε στοιχεία. Έχουμε λοιπόν 16 ε, μονάδες των Ηνωμένων Εθνών που ε, αναλαμβάνουν την έκθεση για το Γενικό Γραμματέα. Μετά έχουμε άλλη μια έκθεση που αφορά τη βιωσιμότητα και τους αναπτυξιακούς στόχους από το 2015 και μετά όπως τις έχουν περιγράψει οι ε, επιχειρήσεις που έχουν προσχωρήσει στην προσπάθεια αυτή των Εθνών. Η έκθεση λοιπόν αυτή της ομάδας ψηλοεπιπέδου είναι μία σημαντική συμβολή αλλά όχι η μοναδική στην έκθεση που θα υποβάλει στις 25 Σεπτεμβρίου στη Γενική Συνέλευση ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Και πριν να υπογραμμίσω κάποια στοιχεία της εκθέσεως περιγράφοντάς τα, επιτρέψτε μου να πω που βρισκόμαστε τώρα το το 2013 σε σχέση με τους στόχους της χιλιετίας. Θα έλεγα ότι το ποτήρι λοιπόν είναι κάπως περισσότερο από ό,τι μισογεμάτο. Τα 700 εκατομμύρια των ε, πολιτών που βγήκαν από τη φτώχεια και μειώθηκε έτσι από το 2010 ήδη από το 47% στο 22% το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν στην ε, ε, φτώχεια, αλλά και η βελτίωση των υδάτινων ε, πόρων κατά τρόπο ώστε 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, ή ε, τα ποσοστά επίσης της θνησιμότητας, της ελονοσίας, της ε, έχουν μειωθεί με βάση τους στόχους και έχουν ικανοποιηθεί οι στόχοι. Και μπορούμε να πούμε ότι έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα ποσοστά στα στόχους αυτούς. Η μείωση της πείνας μπορεί να μην έχει επιτευχθεί ακόμη, αλλά το 2015 μάλλον θα έχουμε αγγίξει τους στόχους, γιατί ο δείκτης αυτή τη στιγμή είναι μείωση από το 23% στο 14%. Τα καταφέρουμε ακόμα, πιστεύουμε. Πάντως πρόκειται μόνο για στόχους που είχαμε ορίσει στο 2015 και η έκθεση των ε, εταίρων ψηλού επίπεδου μας υπενθυμίζει ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε κανέναν ε, στο περιθώριο. Δηλαδή δεν μπορούμε να δεχθούμε μισή φτώχεια ή μισή πείνα. Όλη η ανθρωπότητα έχει δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή διαβίωση. Η έκθεση λοιπόν αυτή της ομάδας υψηλού επίπεδου λαμβάνει υπόψη νέε παραμέτρους, παραμέτρους που δεν είχαμε στη διάθεσή μας όταν ξεκίνησε αυτή η πρώτη προσπάθεια, όπως οι κλιματικές αλλαγές, η επιταχυνούμενη αστιφιλία, οι αυξανόμενες ε, ε, ανισότητες μέσα στις χώρες, το η τη αύξηση της ανεργίας και κυρίως των νέων και από την άλλη η νέα και παγκόσμια συνθεσιμότητα και ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην παγκοσμιοποίηση, δημογραφικές τάσεις, κατανάλωση, τα μοντέλα κατανάλωσης και παραγωγής και εδώ βλέπουμε ότι χρειάζεται μια παγκόσμια, ένα παγκόσμιο θεματολόγιο και ένα παγκόσμιο οικουμενικό πλαίσιο που θα ισχύει για τους πάντες, έστω και αν οι στόχοι μπορούν για την κάθε χώρα να περιγραφούν με πιο συγκεκριμένους όρους. Άρα έχουμε πέντε μεταλλακτικές τροποποιήσεις που χρειάζονται. Ε, η πρώτη είναι αυτή που αναφέρει μόλις τώρα ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε κανένα στο περιθώριο. η δεύτερη μεταλλακτική τροποποίηση είναι η βιωσιμότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη να μπουν στο πλαίσιο, να μπουν στο επίκεντρο μάλλον του πλαισίου της ε, ανάπτυξης. Η ανάπτυξη και η ε, συμπεριληπτική ε, απασχόληση για την καταπολέμηση της ανεργίας και μια νέα παγκόσμια εταιρική σχέση. Η ομάδα εργασίας η ομάδα υψηλού επίπεδου έχει θεσπίσει αρχές και στόχους περισσότερο και όχι, δεν έχει περιγράψει λεπτομέρως τι θα πρέπει να ε, συμβεί για να επιτευχθεί ο κάθε στόχος ή τους όρους αυτού. Αλλά πάντως επιβεβαιώνει και την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενθαρρύνει η ομάδα υψηλού επίπεδου το ενιαίο πλαίσιο με στόχους και ε, αποτελέσματα που χωρίζονται να δεσμευτικά μπορούν να αποτελέσουν ένα μέτρο σύγκρισης και, παρα... και επιτήρησης της υλοποίησης. Και επίσης, εάν θέλουμε να παρακολουθούμε σοβαρότητα την κατάσταση και μπορούν να μας προσφέρουν τις λεπτομέρειες για την καταπολέμηση παραδείγματι των ισοτήτων στην πρόσβαση παραδείγματι, οι στόχοι θα πρέπει να θεσπιστούν σε εθνικό επίπεδο και θα πρέπει να θεωρηθεί ότι μόνο όταν, τηρούν, όταν έχουν πληρωθεί μάλλον για κάθε σχετική ομάδα ε, πληθυσμού ή εισοδήματος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πιστεύω κατά τη δική μου γνώμη. Έμεσα δηλαδή αυτή η προϋπόθεση καλύπτει το ζήτημα της ανισότητας. Ο κάθε στόχος θεωρείται ότι πληρείται μόνο όταν έχει εκπληρώσει το ποσοστό που απαιτείται για το κάθε κομμάτι του πληθυσμού και έτσι δεν αφήνουμε κανένα να χαθεί μέσα από αυτή την καταδυνάστευση των μέσων όρων που μπορεί να παραλλάξουν σημαντικά την κατάσταση και να τη δείξουν πολύ πιο ρόδιμη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Και έτσι ε, δεν αναφερόμαστε μόνο σε παρακολούθηση των μέσων όρων, αλλά σε ανάλυση της στήριξης των προϋποθέσεων και των στόχων για κάθε κομμάτι της κοινωνίας. Τώρα, θα ήταν ίσως περιβολικά λαζονικό το να πούμε δύο χρόνια πριν ε, την, ποιοι θα έπρεπε να είναι οι στόχοι που θα υλοποιηθούν το 2015. Γι' αυτό λοιπόν εμείς απλώς περιγράφουμε όχι ένα σενάριο, αλλά μια γενική εικόνα, μια ιδέα και ένα πλαίσιο Ένα παράδειγμα σχετικά ε, πλήρες, γιατί ουσιαστικά ακολουθεί το υφιστάμενο πλαίσιο, αλλά συμπληρώνει και νέα στοιχεία, την ενέργεια της εργασίας, ε, την ειρήνη και ασφάλεια την ε, χρηστή διακυβέρνηση, στοιχεία δηλαδή τα οποία αποτελούν ε, συμπλήρωμα, ε, χάρη, συμπληρώνουν χάρη στις παλαιότερες επικρίσεις που είχαν διατυπωθεί, τις παλαιές αρχές και αξίες. Δεν μπορεί βέβαια αυτή η έκθεση να θεωρηθεί το τέρμα μιας διαδικασίας. Επί παραδείγματι χρειάζεται να διευκρινιστεί περαιπέτερο τι είδου μορφή μπορεί να αναλάβει για, την για το αναπτυξιακό αυτό πλαίσιο η εταιρική σχέση και μπορεί να οδηγήσει σε μια περαιτέρω συζήτηση για το αν η ανάπτυξη, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων, όχι μόνο στο εισόδημα, αλλά και σε ευκαιρίες, μεταφορές και το καθεξής, μπορεί να αποτελέσει έναν σκοπό και πώς μπορεί αυτός να υλοποιηθεί. Για να επιτευχθεί η ισότητα ευκαιριών, επίσης η ομάδα προτείνει την ανάλυση των δεδομένων προτιμένου να επαληθεύεται ότι για κάθε κατηγορία πληθυσμού πληρούνται οι στόχοι. Και τα τελευταία δύο σημεία που καλύπτουμε έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση. όπου γίνεται πρόταση για ένα ενιαίο πλαίσιο με την ροή πόρων που θα παράγονται από τη βιωσιμότητα, από την πράσινη ανάπτυξη, τα λεγόμενα πράσινα κονδύλια που θα έχουν συνοχή σε σχέση με το αναπτυξιακό πλαίσιο. Ιδάλλως δεν έχει νόημα να, επιδιώκουμε ένα ενιαίο αναπτυξιακό πλαίσιο και στη συνέχεια να το υπονομεύουμε με διάχυση των πόρων ή με εσφαλμένη χρήση τους. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει μια ενιαία πηγή σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση αυτού του πλαισίου, όποιο είναι, και μια ενιαία διαδικασία παραγωγής έκθεσης για, την, ε, για τις προοπτικές της ενιαίας παγκόσμιας ανάπτυξης που θα υποβάλλεται κάθε χρόνο. Όπως είπε, η διαδικασία δεν έχει κλείσει, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Η έρευνα που συνεχίζεται επιγραμμικά με επισκέψη, επισκέψη πάνω από ενός εκατομμυρίου ενδιαφερομένων δίνει εντυπωσιακά και ενδιαφέροντα πολλές φορές ε, αποτελέσματα ότι η διαφάνεια παραδείγματι και η χρηστή διακυβέρνηση μετά την εκπαίδευση και την υγεία θεωρείται τρίτη αξία ε, από τους επισκέπτες που μέσω του διαδικτύου καταθέτουν τις απόψεις τους και θα πρέπει να πάρει μεγάλη και υψηλή θέση σε αυτό το πλαίσιο. Οι διαβουλεύσεις αυτές συνεχίζονται σε επίπεδο κρατών στο τέλος της διαδικασίας θα έχουν αναπτύξει τις εθνικές διαβουλεύσεις πάνω από, 1000, από 100 χώρες και είναι ενδιαφέρουσα αυτή η διαβούλευση γιατί έχουμε να κάνουμε διάφορες ομάδες πληθυσμού και ηλικιακές αλλά και επαγγελματικέ. Ενισχύεται έτσι η κατεύθυνση με τις πολιτικές που έχει χαράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που πιστεύω ότι είναι συμβατές και συνεπείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα προχωρεί περισσότερο από ό,τι έκθεση και ζητάει την συνοχή της στην ανάπτυξη. Εάν σκεφτούμε ότι μια νέο πλαίσιο, μια συντονισμένη ροή των πόρων, ένα εφαρμοζόμενο, ένα σωστά εφαρμοζόμενο πλαίσιο και η ανάγκη του συντονισμού σε κάθε πλαίσιο και διεθνώς της συνοχής, όταν μάλιστα δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί και δεν έχουν ρονταριστεί οι σχετικοί μηχανισμοί. Πρέπει πλέον, ύστερα από την ε, στα λόγια αναφορά σε τόσες πολλές εκθέσεις να περάσει στην υλοποίηση γιατί χρειάζεται να υπάρχει το πλαίσιο. Τα συμπέρασμα λοιπόν, τα συμπεράσματα για να προχωρήσουμε πέραν της ανάπτυξης και της ε, προόδου που αναφέρεται στα τελευταία ψηφίσματα μπορεί να ε, υπογραμμίσετε λιγότερο στο έγχρο της ομάδα εργασία, αλλά θα πρέπει να επιδιωχθεί, γιατί όταν μιλούμε για μηδενική φτώχεια, μηδενική πείνα έως το 2030, θα πρέπει και να πούμε προκαταβολικά εάν μας φαίνεται ικανοποιητική ως επίπεδο ε, ικανοποιητικό το επίπεδο της φτώχειας με 1,25 δολάρια την ημέρα ή αν θέλουμε να κάνουμε προσπάθεια για περισσότερη μείωσή τη. Αλλά πρέπει και αυτό να το παρακολουθούμε και να το επαληθεύουμε. Βεβαίως ε, υπάρχει πρόταση για υιοθέτηση και των εθνικών γραμμών φτώχειας πέραν του μέτρου σύγκρισης κρίσεως της φτώχειας. Ευχαριστώ πολύ. Merci Σας ευχαριστούμε. Θα σας δώσουμε 15 λεπτά για τους τρεις ομιλητές. Μπορείτε να κατανείμουμε το χρόνο όπως επιθυμείτε. Ο κύριος Μέγερς. Εντάξει, θα αρχίσω εγώ και θα συμπληρώσουμε κάποια στοιχεία οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι προβλέπετε ως προς ε, τις πολιτικές εκδηλώσεις και διαδικασίες από πλευρά σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η ΕΕ και το Κοινοβούλιο να συνεργαστούν στενότερα ούτως ώστε η επιρροή τους να μεγεθυνθεί ε, μετά από την εφαρμογή του νέου πλαισίου της πολιτικής μας για την περίοδο μετά το 2015. Θα ήθελα να σας ε, δώσω κάποιες πρώτες εντυπώσεις για την ετήσια έκθεση και οι συνάδελφοι θα σχολιάσουν τις ε, λεπτομέρειες και τις βασικές αρχές. Εν γέννη λοιπόν, παρότι το είπατε ήδη, θα λέγαμε ότι υπάρχουν ε, διαφορετικές ε, μικτές αντιδράσεις από πλευράς με κυβερνητικών οργανώσεων, όμως Εν γέννη ήταν πιο ικανοποιητική η έκθεση από ό,τι περιμέναμε, ε, όχι από όσο ελπίζαμε, αλλά από όσο περιμέναμε. Ε, ε, στο Μπάλι στη σύσκεψη της ομάδας ε, υψηλού επίπεδου δύο μέρες μετά την βασική σύσκεψη συναντηθήκαμε με τους αρμοδίους για τη σύνταξη της έκθεσης και η επισκόπηση που μας έκανε των αντιδράσεων των εκπροσώπων 250 μη κυβερνητικών οργανώσεων ήταν μάλλον απογοητευτική και ήταν πολύ υπό τον προσδοκιών μας. Ε, σε αυτή λοιπόν την ε, συνάντηση υπήρξαν νέες αντιδράσεις από πλευράς μας και από πλευράς ε, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και όλων των εμπλεκομένων σε αυτό το πάνελ υψηλού επίπεδου για να αυξήσουμε τις προσδοκίες και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Βοήθησε λοιπόν αυτό από ό,τι φαίνεται. Είναι μεγάλο το δυναμικό του κειμένου. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και για κάποια ζητήματα είναι αρκετά ισχυρή η φραζολογία που χρησιμοποιείται. πάντω. Ε, το γενικότερο αίσθημα ήταν αυτό τη ανακούφιση όταν είδαμε ε, την έκθεση. Παρ' όλα αυτά παραμένουμε σε μια κατάσταση όπου ανησυχούμε διότι ε, διαπιστώνεται διαβάζοντας το έγγραφο ότι θα αποτελέσει μια, ένα χάρτη για το μέλλον, ένα οδικό χάρτη για τα επόμενα 20 χρόνια. Ε, όμως ε, υπάρχουν και φράσεις που έχουν αντιγραφεί από προηγούμενες εκδηλώσεις ε, και έγγραφα και δηλώσεις και φαίνεται σαν ένα στάνταρ κείμενο του ΟΗΕ. Ε, και θα κυκλοφορήσουν πολλά τέτοια έγγραφα το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τις αρχές του κειμένου αλλά νομίζω ότι σίγουρα δεν θα αποτελέσει τελικά αυτό το έγγραφο τον οδικό χάρτη για το μέλλον διότι παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες ακριβώς λόγω του ότι αντιγράφονται τμήματα από προηγούμενες δηλώσεις δεν επαρκεί ε, το να βρούμε μια καλύτερη διατύπωση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ουσία. Ψαχνώ να πούν ακριβώς ε, τι εννοούν. Όλοι χρησιμοποιούμε μια τυποποιημένη ε, καθολι καθο... φρασολογία, καθολικότητα, βιωσιμότητα και όλα τα σεότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε την ουσία λογοδοσία παραδείγματο χάρη. Ναι, για, την εξετάζουμε σε τοπικό επίπεδο, αλλά δεν λέμε τίποτα για το διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο η διαδικασία και τα όλα όσα θα συμβούν σε επόμενες εβδομάδες και μήνες θα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Όπως είπε μόλις τώρα ο κύριος Βιτζιλάντη, Βάσει της αρχής ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανείς εμέσως ε, πραγματευόμαστε το θέμα των ανισοτήτων ε, προς το παρόν. Δυστυχώς. Πολλά θα εξαρτηθούν ε, από, την, από τον ανασχηματισμό του κειμένου της επόμενης εβδομάδας για να χρησιμοποιηθεί τον έγγραφο στις διαπραγματεύσει, Θα ακούσουμε όμως παρόλα αυτά του συναδέλφου να μα μιλάνε για κάποιε βασικές αρχές που διέπουν το κείμενο. Ευχαριστούμε κυρία Σαλντάνια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα στην αρχή να σας πω, όπως ανέφερε και ο κύριος Βιτζιλάντη, ότι εμείς οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών ε, καλωσορίζουμε την αύξηση των διαβουλεύσεων και της συμμετοχικής διαδικασίας που επικράτησε για τη σύνταξη ε, του εγγράφου. Βεβαίως μετά από όλες τις επενδύσεις που κάναμε εμείς ε, από πλευράς χρόνου και ενέργειας απογοητευτήκαμε από το πόνημα, το τελικό πόνημα και όπως είπατε και εσείς είναι ανάμεικτα τα αισθήματα κυριαρχεί η αρνητική εικόνα, προσπαθούμε να κεντρωνόμαστε στα θετικά σημεία. Ξέρουμε ότι είναι μια ε, δύσκολη διαπραγματευτική διαδικασία. Ελπίζουμε να συνασπιστούμε, ώστε ε, να μπορέσουμε να προωθήσουμε τουλάχιστον ε, τις θετικές πτυχές της έκθεσης και να μην επικρατήσουν τα αρνητικά σημεία στο δημόσιο διάλογο. Όπως ακούσαμε και νωρίτερα, η πρώτη αλλαγή που αναφέρεται ως στόχος και είναι ένα από τα βασικότερα μηνύματα του κειμένου πρέπει να ληφθεί υπόψη στις μελλοντικές συζητήσεις, διότι προκρίνεται μια προσέγγιση κοντά στη ρίζα. Αυτό ζητάει η κοινωνία των πολιτών, να μην ασχολούμαστε μόνο με τα συμπτώματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά να δούμε τις δομές, τις υποδομές και τις διαδικασίες που γεννούν την φτώχεια. Ε, στη συνέχεια να αναγνωριστεί ότι η φτώχεια προέρχεται από ένα σύνολο παραγόντων που συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και έτσι πρέπει να προσεγγίζουμε το πρόβλημα ε, της φτώχειας. Ε, στείλαμε για Λάβαμε την περασμένη εβδομάδα μια ανοιχτή επιστολή από τον το αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον ΟΗΕ και ζητούμε να ληφθεί σοβαρά υπόψη αυτή η επιστολή για τις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις και συζητήσεις για την ατζέντα μετά το 2015 μπορεί δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μια πλούστατη εξίσωση που να σχετίζεται μόνο με το εισόδημα για να οριοθετήσουμε την φτώχεια. Δεν μιλάμε για το 1,25 δολάρια την ημέρα. Είναι ε, υπερβολικά μινιμαλιστικός αυτός ο στόχος. Δεύτερον, η ισότητα και μη διακριτική μεταχείριση, βασικές έννοιες στις οποίες αναφέρθηκα και νωρίτερα, η επιταγή της καταπολέμησης ανισότητας έχει τρεις διαστάσεις. Υπάρχει η ισότητα, δηλαδή ίσες ευκαιρίες και ίσα ωφέλη. Στη συνέχεια η ανισότητα και η διακριτική μεταχείριση. Αυτές, αυτά είναι τα τρία σκέλη της προσπάθειας που γίνεται για την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Προτείνεται μια οριζόντια, εγκάρσια προσέγγιση ε, μιλάμε για την άρση των φραγμών, για την πρόσβαση σε ζωτική σημασία υπηρεσίες. Αναφερόμαστε σε συγκεκριμένους στόχους για την πρόσβαση σε υπηρεσίες δικαιοσύνη, παραδείγματο χάρη, και ε, ομαδοποίηση των μέτρων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το τομέα. Όπως είπε και ο συνάδελφος όμως, η ανισότητα ε, είναι κάτι που χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία. Υπάρχουν κοινωνικά μηνύματα, λαϊκές εξεγέρσεις κατά της ανισότητας ανά τον κόσμο και είναι κρίμα, πιστεύουμε, που δεν απηχείται αυτό μέσα στην έκθεση το, η μία αναγνώριση αυτού του φαινομένου από την έκθεση μας οδηγεί σε μία γκρίζα ζώνη τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς όμως να δίνουμε συγκεκριμένες ε, ιδέες για το πώς θα επιτευχθεί αυτό. Επίσης ε, υπάρχει ατζέντα του αξιοπρεπούς κόσμου η οποία τελικά δεν συμπεριληφθήκε ε, ο, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ε, θεωρεί ότι αυτό είναι υπερβολικά φιλόδοξο για τις αναπτυσσόμενες χώρες και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν συμπεριλήφθηκε. Εμείς όμως θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένους στόχους για τις ίσες ευκαιρίες και να μην ε, περιοριζόμαστε ε, σε κάποιες επιτυχές π.χ. της ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλλα ε, κινητοποίηση των μέσων φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή σε σχέση με τον στόχο 12 είναι μια σειρά από συνιστός αυτής της ατζέντα που πρέπει να συμπεριληφθούν οπωσδήποτε μέσα στο έγγραφο κατόπιν. Καλωσορίζουμε το θέμα της ε, περιβαλλοντικής ε, λογοδοσίας ε, σε σχέση με την αηφόρο ανάπτυξη. Αφ, ε, χαιρόμαστε που τελικά συμπεριλήφθη, αλλά όμως λείπουν άλλα σημεία, όπως η αξιοπρεπής εργασία. Η έκθεση κάνει πολύ περιορισμένες συστάσεις για συγκεκριμένο τρόπο δράσης ε, για τα χρόνια μετά το 2015. Δεν μιλάει για το παγκόσμιο πλαίσιο και ως προς τις κλιματικές αλλαγές και την ευθύνη των ε, αναπτυσσόμενων χωρών για την ε, παραγωγή και την κατανάλωση, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχουν πιο συγκεκριμένα στοιχεία και διαφοροποίηση της ευθύνης που αποδίδεται. Ε, και ε, κυρίως να συμπεριληφθούν και οι μηχανισμοί λογοδοσίας ε, που είχαν προβλεφθεί στην αρχή σε σχέση με τους στόχους της χιλιετίας. Ποιοι είναι οι κάτοχοι των δικαιωμάτων, ποιοι είναι υπεύθυνοι για τα τέλη, για κάθε εντεταλμένη δράση και για κάθε οργανισμό, περνώντας από το τοπικό επίπεδο στο εθνικό και το διεθνές, να είναι ξεκάθαρες οι ευθύνες, να είναι ξεκάθαρο σε ποιον λογοδοτούν και επίσης εφαρμοσιμότητα ε, των στόχων ε, που τίθενται. Νομίζουμε ότι αυτό είναι κέρια σημασίας και γι' αυτό ε, θεωρούμε ότι το πλαίσιο μετά το 2015 θα αποτύχει αν δεν υπάρχει το στοιχείο της λογοδοσίας. Είναι βασικός πυλώνας των συζητήσεων που γίνονται για το αναπτυξιακό πλαίσιο μετά το 2015. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Βάντερς τώρα. Θα σεβαστώ ελπίζω το χρόνο. Ο συνάδελφος υπογράμισε θα έλεγα. κάποια προβλήματα τα οποία παρουσιάζει η εργασία κάποιων ιδιαίτερα ικανών και αποτελεσματικών ανθρώπων. Οι γνώμες πάντως προέρχονται από 2.000 μικιό. Το δικό μας έγγραφο, το οποίο εμείς έχουμε, έχει τον τίτλο τον λίγο φοβιστικό ότι πρέπει οι άνθρωποι να πάρουν την πρώτη θέση, ο πλανήτης την πρώτη θέση και δεν μπορούμε πια να λέμε business as usual. Πρέπει να υπάρχει, ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να εκφράσουμε την άποψή μας σε αυτή τη συνάντηση και ελπίζω να είναι αρχή ενός καλύτερου και πιο μόνιμου διαλόγου ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών. Ε, η κοινωνία των πολιτών εκπροσωπεί τους πολίτες τους οποίους εκπροσωπεί και το Κοινοβούλιο. Τα θέματα αυτά έχουν την ίδια σημασία για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και για τους πολίτες όλου του πλανήτη. Δεν μπορούμε λοιπόν να περιοριστούμε στους παραδοσιακούς εταίρους ε, της ανάπτυξης και να περιοριστούμε στο ε, παράδειγμα, το, ε, σε εισαγωγικά παράδειγμα που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα τον προηγούμενο αιώνα και την πρώτη δεκαετία ίσως ε, του αιώνα μας. Σχετικά τώρα με τις αποφάσεις το Σεπτέμβριο της πιθανές στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ελπίζουμε οδεύοντας προς το συμβάν αυτό να μπορέσουμε να καταλήξουμε και να συμφωνήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις βασικές αρχές της έκθεσης υψηλού επίπεδου που θα πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστές τώρα που η διαδικασία μετατρέπεται περισσότερο σε διαδικασία cut and paste διακυβερνητικού τύπου. Οι εργασίες της ανοιχτής ομάδας εργασίας θα ακολουθήσει μετά την ε, συνέλευση του Σεπτεμβρίου μέχρι το τέλος του 2014. Ελπίζουμε ότι η κοινωνία των πολιτών θα μπορέσει να συνεισφέρει και να αποτελέσει και τμήμα ίσως της αντιπροσωπείας που θα επισκεφθεί την Νέα Υόρκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εμπειρία αυτή θα συνεχιστεί για την οποία σας είμαι θα ευγνώμονες και το 14 και το 15 που είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ανησυχίες που εκφράσατε. Κύριε Γκέρενς, έχετε ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε καταλήγουμε στο τέλος μιας σειράς πολύ ενδιαφέρουσων παρουσιάσεων. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο όμως για το θέμα της διακυβέρνησης. Ποιος κάνει τι και ποιος είναι υπεύθυνος γιατί. Ποιος θα είναι ο ρόλος των κυβερνήσεων, ποιος θα είναι ο ρόλος των ΜΚΟ, μπορείτε να αναπτύξετε λίγο περισσότερο το συγκεκριμένο θέμα. Γνωρίζουμε ότι οι λεγόμενοι παραδοσιακοί ε, πρωταγωνιστές της διαδικασίας αυτές είναι τα κράτη-μέλη, είναι η Ένωση, οι διεθνείς οργανισμοί. Αλλά εδώ από το τέλος του ψυχρού πολέμου και μετά και ιδιαίτερα μετά από, το, από τη φάση στα πλαίσια της οποίας άρχισαν να αναφέρονται και νέοι εταίροι όπως στη Συμφωνία του Κοτονού, ο ιδιωτικός τομέας, η ΜΚΙΟ, παίζουν και αυτοί ένα σημαντικότατο ρόλο. Θα ήθελα λοιπόν να με διαφωτίσετε λίγο ε, γύρω από τις προοπτικές τις οποίες εσείς ανοίγετε. Τι μπορούμε να κάνουμε για την πρόθεση λοιπόν μιας καλύτερης διακυβέρνησης. Ένα παράδειγμα, σε κάποιες χώρες δεν λειτουργεί τίποτα. Η ένδυα είναι σχεδόν ενδυμική. Η σωστή διακυβέρνηση λείπει και είμαστε ανίκανοι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν κράτη-μέλη να δημιουργήσουμε πραγματικούς χώρους συνεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, σαν παράδειγμα, ποιος θα είναι ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Γιατί επαναλαμβάνω ότι τα κράτη έχουν εξαντλήσει τα όρια τους θα μπορέσατε σαν παράδειγμα να σκεφτείτε κάποιους θεσμικούς εταίρους που διαπραγματεύονται ένα χώρο συνεργασίας στο εσωτερικό αυτών των χωρών. Έτσι ώστε να υπάρξει χώρος και για τις μη κρατικέ ε, οργανώσεις που θα μπορούσαν να δράσουν σε ένα πλαίσιο ε, ε, δεοντολογικά αυστηρότατο. Ένα παράδειγμα ήταν αυτό το οποίο μπορεί να ανοίξει αυτή τη συζήτηση για τη διακυβέρνηση. Σας ευχαριστώ κύριε Γκέρεντς. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Μπέρμαν. Για τη νέα έκθεση για την ανάπτυξη μετά το 2015. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μια ερώτηση για το Vigilante. Ευχαριστώ για την έκθεσή σας, την οποία λυπάμαι αλλά δεν διάβασα ακόμα. Συγγνώμη γι' αυτό. Όταν πριν μερικούς μήνες μας επισκέφθηκε η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Στα πλαίσια της συζήτησης αυτή φάνηκε ότι στην υπηρεσία την αναπτυξιακή του ΟΗΕ υπάρχουν ανησυχίε σχετικά με την προάσπιση της καθολικότητας των αξιών. υπόθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει έναν ρόλο εκπροσώπου αυτών που υπερασπίζονται αυτές τις καθολικές αξίες. Πώς βλέπετε τη συζήτηση αυτή. Είσαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η συζήτηση μέχρι σήμερα ή μήπως ανησυχείτε όσο ανησυχούσατε και στο παρελθόν. Πριν σας ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Βιτζιλάντε και στα μέλη του πάνελ, ε, θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Γκασπάρ Φαντινή έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω κάποια σχόλια και να παρουσιάσω απόψε Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτήν τόσο σημαντική έκθεση της ομάδας ψηλού επίπεδου. Οι περισσότεροι θα γνωρίζετε ότι ο Επίτροπος Πίμπαλξ ήταν ένα από τα μέλη της Επιτροπής αυτής και μετήχε εκτεταμένα στις εργασίες του πάνελ. Ο Επίτροπος Πίμπαλξ είναι αρκετά ικανοποιημένος με την έκβαση των εργασιών της ομάδας και το του στην έκθεση. Ε, σίγουρα δεν είναι το τέλος της διαδικασίας, ε, όμως θεωρούμε ότι συνιστά ένα πολύ σημαντικό στοιχείο μεταξύ άλλων στοιχείων που θα μας συνοδεύσουν να ε, εισέλθουμε στο πλαίσιο post 2015. Βλέπουμε ξεκάθαρους προσανατολισμούς και προτεραιότητες από πλευράς ε, αυτού του πάνελ ε, που ε, συνάδουν με τα τις δικές μας συστάσεις της ανακοίνωσεις μας και τα αυριανά συμπεράσματα του Συμβουλίου κατά πάσα πιθανότητα. θέλουμε να έχουμε μια ενιαία ατζέντα και οι ανησυχίες που έχουμε για την κατάργηση της φτώγειας να συνδυαστούν με τις προσπάθειές μας για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης πρέπει να είναι καθολικό αυτό το θεματολόγιο, είναι σημαντικό για όλες τις χώρες, ε, στο μέτρο που θέλουμε ε, πραγματικά να μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη. Στη συνέχεια, η έμφαση δόθη στο θέμα της ε, καταπολέμησης των ανισοτήτων, επίτευξη της ε, ισότητας είναι ένα διαρκής ε, προβληματισμός. Επίσης το θέμα του κράτους δικαίου, η ασφάλεια και η ειρήνη και το ειδικό βάρος που έχουν. Ξαναλέω ότι όλες οι στάσεις Επιτροπής συνάδουμε με τις δικές μας σε αυτά τα ζητήματα. Όπως μας εξήγησε ο κύριος Βιτζιλάντε, η έκθεση του πάνελ υψηλού επίπεδου μας μιλάει για πέντε διαρθωτικού χαρακτήρα καμπές ε, ε, δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, η βιώσιμη ανάπτυξη, η αλληλέγγυα ανάπτυξη, ε, λογοδοσία για όλους και νέα παγκόσμια εταιρική σχέση πέμπτον. Εάν δείτε ε, τα πέντε δομικά στοιχεία της ανακοίνωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα διαπιστώσετε μεγάλη σύγκληση σε σχέση με αυτούς τους πέντε στόχους, τουλάχιστον με τους τέσσερις πρώτους στόχους ε, αξιοπρεπή σε συνθήκες διαβίωσης, ε, βιώσιμη ανάπτυξη, καλή διαχείριση των φυσικών πόρων. Είναι πράγματα που προτείνουμε και εμείς και με ποιο τρόπο κράτος δικαίου, καλή διακυβέρνηση, σεβασμός ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ξεχωριστός στόχος ε, για την ασφάλεια και την ειρήνη, το πάνελ ενσωμάτωσε αυτούς τους δύο διακριτούς στόχους σε έναν, αλλά δεν υπάρχει κάποια αντίφαση. Το, το πάνελ επίσης εν είδη παραδείγματος θέτει το ένα δωδεκάλογο, 12 στόχους είναι σημαντικό όμως να ε, διευκρινίσουμε ότι παρότι δεν πρόκειται για τελικούς στόχους, ε, είναι εφικτά αυτά που επιδιώκουν αμφότερες οι πλευρές, διότι ακριβώς δεν υπάρχουν αντιφάσεις ανάμεσα στο πόρισμα του πάνελ και την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ σημαντικό αυτό. Εξίσου σημαντικό είναι να πούμε ότι παρότι ε, το πάνελ συναποτελείται από ανθρώπους που δεν ε, ήταν εκεί με την προσωπική τους ιδιότητα, εκπροσωπούσαν ε, φορείς ε, και οργανισμούς και όμως προέρχονταν από 27 διαφορετικά background και άρα ακούστηκαν πολλές διαφορετικές φωνές στις εργασίες αυτού του πάνελ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, και θα συμβάλλει στο γενικότερο προβληματισμό μας για την κατάσταση μετά το 2015. Ευχαριστούμε. Θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Βιτζιλάντη για να απαντήσει και για να κάνει καταληκτικές ε, παρατηρήσεις. Ε, πρώτον, να ξεκαθαρίσω ότι πρόκειται για μια έκθεση που υποβάλλουμε στο Γενικό Γραμματέα. Δεν είναι έκθεση του ΟΗΕ. Είναι μια έκθεση που θα χρησιμοποιήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για να κάνει τη δική του υποβολή αναφοράς προς τα κράτη-μέλη το Σεπτέμβρη. Ε, σας είπα ότι ο εταιρικός κόσμος, ο ιδιωτικός τομέας και οι εταιρείε που έχουν προσπογράψει το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ θα στείλουν τη συνεισφορά τους και 60 διαφορετικοί οργανισμοί του ΟΗΕ που συντονίζουν τη δράση τους στα πλαίσια μιας ειδική ομάδας δράσης που έχει ήδη συντάξει με έκθεση. Επίσης θα συμβάλλουν στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Λοιπόν, ε, η ανισότητα όντω την προσεγγίζουμε εμέσω μέσα στην έκθεση. Αληθεύει αυτό, διότι ε, όταν μιλάμε για την μέτρηση και την ανάλυση των στατιστικών αποτελεσμάτων. Ε, πιστεύουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά πιστεύω σε κάθε περίπτωση ότι δύσκολα μπορούμε να καταλήξουμε συμφωνία για ένα στόχο καταπολέμησης ε, της ανισότητας. Εύκολα μπορούμε να μιλήσουμε για καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες και να συμφωνήσουμε για ένα συγκεκριμένο στόχο. Εύκολα σε επίπεδο διεθνούς ε, κοινότητα μπορούμε να μιλήσουμε για διεθνή προστασία, μπορούμε να συμφωνήσουμε για την ισότητα των ευκαιριών. Ναι, αλλά για τι εισοδηματικέ διαφορέ, ε, το να θέσουμε ένα φιλόδοξο στόχο, ιδεολογικό πώ παρουσιάζει μεγάλε δυσκολίε. Πιστεύω λοιπόν ότι η μοναδική διατύπωση που θα ήταν ε, πιθανή για τέτοιου είδου πάνελ θα ήταν να μειώσουμε εν γέννη τι ανισότητε. Μέχρι πού όμω, το 0% είναι ουτοπία. Ε, και αν ανέβουμε προς την άλλη κατεύθυνση είναι αυθαίρετο. Καταλαβαίνετε, ξεκινάει μια κάπως φιλοσοφική συζήτηση σε σχέση με το στόχο ε, για το εισόδημα ως προς τις ανισότητες και θα πρέπει να κατευθυνθούμε προς ε, ποιο στόχο ακριβώς, καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες, προστασία για όλους κτλ. Εδώ θέτω ένα μάλλον ρητορικό ερώτημα, δεν έχω συγκεκριμένη απάντηση. Αυτό εξηγεί όμως γιατί το πάνελ ε, δεν ε, θέλησε να ε, στοχοθετήσει ως προς την καταπολέμηση των ισοτήτων διότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές πτυχές και αυτό το σλόγγαν, δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι η συνένεση για τους ε, νέους στόχους είναι πιθανή αν επιτευχθεί για κάθε πληθυσμιακή ομάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την καταπολέμηση των ανισοτήτων, ίσως όχι για τις εισοδηματικές ε, ανισότητες, αλλά για όλες τις υπόλοιπες, ε, όσο στον τομέα της υγείας, στον τομέα της συμμετοχής κτλ. Κύριε Μπίρμαν, ε, σε σχέση με το ερώτημά σας, ε, μπορούμε να το συζητήσουμε επί μακρόν, αλλά σε επίπεδο διεθνούς ε, κοινότητας γίνεται μια συζήτηση για τη σχετικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά τη διαστολή με την καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε την παγκόσμια διακήρυξη του 48, αλλά υπάρχουν και δικαιώματα που κυμαίνονται ανα, ανα ήπειρο, ανα χώρα, ομάδα και ούτω καθεξής. Πιστεύουμε ως βασική αξία ότι είναι καθολικά τα δικαιώματα, όμως είναι τελείω απειλεί αυτή η διακήρυξη, αυτή η αρχή. Είναι θεωρητική η απειλή τουλάχιστον θεωρητική. Α δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν τρόποι να επιβεβαιώσουμε την καθολικότητα των δικαιωματών όταν μιλάμε για του στόχου για την ισότητα των δύο και διαβάσετε κάποιε προτάσει και να τονίσω εδώ ότι δεν πρόκειται για τελικούς στόχους χιλιοετίας ε, αναφέρονται εδώ ω ε, εν είδη παραδείγματος. Ε, λέμε για τι γυναίκε ότι θα πρέπει να μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό, να ανοίξουν μια επιχείρηση, να μετέχουν στα κοινά νομίζω ότι είναι αρκετά ισχυρή η διατύπωση για την κατάργηση διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου. Στις συστάσεις του πάνελ θα μπορούσαμε να σας καθησυχάσουμε ως προς κάποιες ανησυχίες που έχετε. Όμως, ε, από πλευράς ε, πρακτικής εφαρμογής σε κάθε χώρα ε, της επιβεβαίωσης αυτών των καθολικών αρχών, εκεί θα πρέπει ε, να εκφράσετε σοβαρότερες ανησυχίες και να σας πω ότι για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξορισμού ανάγεται στο άτομο οποιαδήποτε δήλωση που κάνουμε Και δεν ε, απηχείται αυτό ε, επαρκώς στην έκθεση του πάνελ, αυτό θα το αναγνωρίσω, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν απειλείται λόγω της διατύπωσης η καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Μπίρμεν, ε, κοιτάξτε, Αντώνιο, μιλήσατε για κυβερνήσεις που λογοδοτούν. Accountable governments. Ε, ε, μη αιρετές κυβερνήσεις μπορούν ε, να λογοδοτούν και αυτή είναι η πρώτη ερώτηση και μπορούμε έτσι να παρακάμψουμε το δημοκρατικό έλλειμμα σε κάποιες χώρες μιλώντας για κυβερνήσεις που λογοδοτούν αντί να τονίζουμε ένα από τα βασικότερα οικουμενικά δικαιώματα, το δικαίωμα για μια αιρετή κυβέρνηση. Τι λέτε. σύντομη απάντηση. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μετά, αλλά ε, η εκλογική διαδικασία είναι πολύ σημαντικό βήμα και ε, οι, ξέρετε, ορισμένες ε, μη αιρετές κυβερνήσεις λογοδοτούν πολύ περισσότερο σε σχέση με τις αιρετές. Δεν είναι και εγγύηση, δηλαδή. Απλώς θα έπρεπε να μιλάμε για συμμετοχική δημοκρατία, όπου οι πολίτες επηρεάζουν όχι μόνο τις αποφάσεις ε, και το βίο της χώρας ε, μία φορά στα 4-5 χρόνια, αλλά μιλάμε για ουσιαστική ε, καθημερινή συμμετοχή και επιρροή στα κοινά. Δεν έχουμε στην έκθεση του πάνελ στόχους ε, για να καταργηθούν οι μη αιρετές ε, κυβερνήσεις. Όχι, αυτό δεν αναφέρεται ρητά όμως ε, διαφυλάντως στην αρχή της καλής διακυβέρνησης και εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε, σε ανεξάρτητα ΜΜΕ και συμμετοχή των πολιτών με διαφόρους τρόπους, όπως βλέπετε στο έγγραφο, κατοχυρώνει τη η δημοκρατία. Η πρόεδρος, ε, ε, οι τρεις εκπρόσωποι της Κονκόρτε για δύο λεπτά έκαστος. Ε. Τι γίνεται στις περιπτώσεις χωρών όπου δεν υπάρχει σωστή διακυβέρνηση. Δεν έχουμε κάποια λύση αυτόματη, δεν υπάρχει μηχανή σωστής διακυβέρνησης, αλλά το θέμα είναι αν οι υποδομές και οι διαδικασίες σε τοπικό ή σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο μπορούν να δώσουν, αν θέλετε, στοιχεία ικανοποίηση σχετικά με τον σεβασμό των δικαιωμάτων του πληθυσμού και οικονομικά και πολιτικά και κοινωνικά. Στα πλαίσια της διαδικασίας που οδήγησε στο Ρίο συνήκωση υπήρξε μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή από κάποιους από τους εισηγητές για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα ξεχωριστά δικαιώματα, το δικαίωμα στη διατροφή, στα τρόφιμα, το δικαίωμα στο πόσιμο νερό κτλ. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε τις χάρτες, τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών κάτι το συγκεκριμένο, κάτι το απτό. Και εδώ η κοινωνία των πολιτών έχει να προσφέρει, παίζει έναν παραδοσιακό ρόλο, παρακολουθεί, ελέγχει, καταγγέλει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να τις υποστηρίξουμε. Θα πρέπει επίσης ε, να ενσωματώσουμε σε κάποιες ε, δομές που ε, προετοιμάζουμε τώρα κάποια στοιχεία έτσι ώστε να διευκολύνουμε την πρόσβαση των τοπικών εταίρων να καταγγέλουν τις διαδικασίες όταν πιστεύουν ότι δεν είναι δικές τους σωστές. Ένα λεπτό παρακαλώ. για την ισότητα. Το θέμα είναι τι προτεραιότητα δίδει κανείς. Τώρα η προτεραιότητα δίδεται στην ανάπτυξη και όχι στα θέματα ισότητας. Εμείς σαν κοινωνία των πολιτών προτείνουμε την ισότητα και μιλάμε για τον κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, δηλαδή η ισότητα μπορεί να είναι αυτό που θα αποφασίσει αν θα πετύχει ή θα αποτύχει η συγκεκριμένη προσπάθεια. Αν δεν επιμείνουμε στον τομέα αυτό φοβάμαι ότι δεν θα πετύχουμε την ολοκλήρωση του πλαισίου για το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν δύο πλευρές. Πρώτον, οι τρόποι για τη συμμετοχή στην διατύπωση των πλαισίων και δεύτερον, η συμμετοχή στην ανάπτυξη ε, αυτή καθεαυτή Αυτές δύο διαφορετικές μορφές διατύπωσης θα επιτρέψουν να συνδυάσουμε τις αναπτυξιακές μας προσπάθειες, κάτι το θετικό ε, για τις ομάδες οι οποίες παρεμβαίνουν. Ο συνάδελφος Βάντερς θα ασχοληθεί με τα θέματα της προετοιμασίας για το πλαίσιο. Νομίζω όμως ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το πώς κανονισμοί και κανόνες μπορούν να καταστήσουν ικανό τον ιδιωτικό τομέα να συνεισφέρει περισσότερο στην ανάπτυξη από ό,τι σήμερα. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι πάντα προτεραιότητα του ιδιωτικού τομέα. Αλλά το κοινό καλό είναι προτεραιότητα των κυβερνήσεων και θα πρέπει να δείξουν οι κυβερνήσεις πώς οι προτεραιότητες αυτές μπορεί να ενταχθούν στους κανόνες λειτουργίας τους για να στοχεύουν στην ανάπτυξη κάποια στοιχεία τέθηκαν, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα και αρχές που δεν συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση. Βάντες. Να πω ότι η οργάνωση στην οποία εργάζομαι σε καθημερινή βάση είναι υπερήφανη για αυτά τα οποία συμβαίνουν και γίνονται, αλλά μας φοβίζει λίγο και η εταιρική σχέση που έχουμε συνάψει με μια μεγάλη πολυεθνική χημική εταιρεία έτσι ώστε να βελτιώσουμε την θρεπτική αξία των τροφίμων που παράγονται στις υποανάπτυξη χώρες. Έτσι θα μπορέσουμε, τουλάχιστον αυτό είναι ο βασικός μας φιλόδοξος στόχος, μέσα αυτής της εταιρική σχέσης να αποτρέψουμε την πείνα των παιδιών. Δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει η προσπάθεια. Αυτό που είναι βέβαιο πάντως είναι ότι στο νέο πανόραμα στο οποίο λειτουργούμε πρέπει κανείς να βρει καινοτόμε μορφές χρηματοδότησης γιατί αλλιώς θα καταστούμε όλοι περιττοί. Ευχαριστώ. Γνωρίζετε ότι εμείς θα στείλουμε το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη μια σημαντική αντιπροσωπεία και είμαι βέβαιος ότι η συζήτηση αυτή θα, τροπο, εμπλουτίσει τις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και μοιραστήκατε τις απόψεις σας μαζί μας. Περνάμε τώρα στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να αφήσω την Προεδρία παρακαλώ στον συνάδελφο κύριο Γκέρενς. chers Ας περάσουμε στο σημείο 9 σχετικά με το μίξ επιχορηγήσεων και δανείων για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ 2014-2020. Ε, θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων και ένα briefing από σύσκεψη των πολιτικών ομάδων από τον εισηγητή, τον κύριο Στάζ. Δέκα λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Μετά από έξι χρόνια τεχνικής εργασίας, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια ε, συνεδρίασε στις 21 Ιουνίου την περασμένη Παρασκευή ε, και στις τελευταίες συνεδρίες της Επιτροπής μας είχαμε προετοιμάσει την έκθεση τη θέση μας μάλλον που θα μετέδιδε ο κύριος Μπάρτ Στές ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και των ε, κρατών μελών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. <laughs> Είναι εδώ ο κύριος Στάς. Πολύ καλό αυτό. Πολύ βασικό. Σας δίνω το λόγο για να μας ενημερώσετε ε, για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη. Ευχαριστώ. Ε, Κοίταξε, σε αυτή την Επιτροπή Εργαστήκαμε στο κέντρο Μποχσέτ, ε, συμμετείχαν και τρία μέλη της ε, γραμματείας, εκπροσωπήθηκαν τα κράτη-μέλη, επίσης ε, και δραστηριοποιήθηκαν ε, πάρα πολύ σε αυτό το τομέα. Ε, Προσώπους Παγκόσμιας Τράπεζας, το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης, εγώ δεν ήξερα ότι είχε τράπεζα, το έμαθα και αυτό, και διάφοροι παρατηρητές. Την Παρασκευή συζητήσαμε λοιπόν για τις εργασίες ε, των τεχνικών ομάδων και ε, των προεργασιών που είχαν κάνει. Δεν ήταν όμως μόνο τεχνική συζήτηση, διότι θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια σε σχέση ε, με το στρατηγικό προσανατολισμό που θα ακολουθήσουμε, πέρα από τις τεχνικές συζητήσεις. Τέσσερις βασικές ανησυχίες εξέφρασαν αναφέρθηκαν και στο παρελθόν. Πρώτον, Θα πρέπει να συνδυάσουμε την δράση μας με την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Πολιτική και τον Οκτώβρη στη προηγούμενη συνεδρίαση είπα ότι για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε αυτές τις προτεραιότητες. Ε, στη συνέχεια ανάγκη για διαφάνεια, ενημέρωση του κοινού ε, σε σχέση με τις εξελίξεις ε, η επιλογή των προγραμμάτων, ε, οι χώρες εταίροι των προγραμμάτων, ε, αυξημένη συμμετοχή της κοινωνίας ε, των πολιτών. Κάναμε κάποιες παρατηρήσεις επίσης σε σχέση με την διαχείριση των υποδομών που διαθέτουμε. Αποδυναμώθηκε η συμβολή μας από την στάση κάποιων κρατών μελών που διαρκώς ε, ήγηραν προτάσεις, ε, τις ίδιες προτάσεις ε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Έγινε μια ανταλλαγή απόψεων και ξεκαθαρίστηκε ότι θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η συμβολή του Κοινοβουλίου. Πρόεδρε, δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Θα μπορούσα βεβαίω να επισέλθω και σε λεπτομέρειε ή αν το προτιμάτε, έχω προετοιμάσει ένα έγγραφο με επιμέρου σημεία που προέβαλα εγώ σε αυτή την σύσκεψη και μπορώ να το δώσω στους συναδελφούς. Αποφασίστε και πείτε μου, Πρόεδρε, θέλετε να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, θέλετε να δώσω απλώς το έγγραφο στους συναδέλφους. Επαναλαμβάνω, γαλλιστή, να μπω σε λεπτομέρειες σε σχέση με αυτά που απλώς ε, απαρίθμησα ή ε, ε, αρκεί το προπαρασκευαστικό σημείωμα και τα πρακτικά της συνεδρίασης. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος αν πω σε λεπτομέρειες. Ε, δική σας είναι η απόφαση, Πρόεδρε. Oui, je viens de me concerter maintenant un peu avec l'administration. Euh, je crois que... Λοιπόν, ε, κοιτάω με την ε, γραμματεία. Νομίζω ότι ένα-δύο λεπτά μπορούμε να δώσουμε περιθώριο συζήτηση για τον προπολογισμό. Αλλά είναι τόσο σημαντικό βέβαια το θέμα που οπωσδήποτε πρέπει να μπορέσει να επισέλθεις και στις κατευθυντηρίες γραμμές. Ναι, δέκα σημεία, πολύ σύντομα. Καταρχάς, αυτή αυτό το μέσον ε, σχετίζεται με την ε, συζήτησή μας για το τεχνικό, για τεχνική έκθεση. Είναι για μένα όρος ο μου κάνευ. Δεύτερον, έχω επιμείνει στις ε, λεπτομέρειες γιατί λυπούμε που δίνεται έμφαση στην ενέργεια και τις μεταφορές και λέγεται μόνο ότι θα καταπολεμηθεί η φτώχεια ενώ πρέπει να επιμείνουμε ακόμη περισσότερο στην, στα έργα τα οποία καταπολεμούν τη φτώχεια. Επίσης, μελέτη ε, επιπτώσεων και τέταρτον οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει συστηματικά να συμμετέχουν στην ε, ε, κατάρτιση του κειμένου, αλλά και δραστήρια να εργάζονται έχοντας γνώση της χώρας εταίρου και να συμμετέχουν. Υπάρχουν βέβαια θέματα σε σχέση με την αποδοχή σε τοπικό επίπεδο. Λέγεται ότι θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις που θα πρέπει να είναι βέβαια οικουμενικές, αλλά Ταυτόχρονα και οι κατάλληλοι δείκτες θα πρέπει να ενσωματωθούν τα αποτελέσματα και οι συνέπειες αυτής, αυτού ε, μέσου μείγματος. Επίσης, κάποιοι δείκτες που αναφέρονται μπορούν να ληφθούν ληφθούν υπόψη, να λαμβάνονται υπόψη. Και για τους στόχους της χιλιετίας, διαφοροποίηση βάση φύλου παραδείγματι, πρέπει να είναι ποιοτική, ποσοτική, αποτελεσματική, βιώσιμη οι δείκτες και να καταγράφουν και κοινωνικές συνέπειες και μακροπρόθεσμες συνέπειες. Διαφάνεια και υπευθυνότητα. Και όπως είπαμε, επιμένω ξεκάθαρα να λέγεται ότι η διαφάνεια σημαίνει πως εξηγούμε στην κοινή δικρομή το, την πορεία, τη διαδικασία επιλογής των έργων και επαληθεύουμε όταν ένα έργο έχει επιλεγεί στην εκτέλεσή του με τα πρακτικά τα οποία είναι, διαθέσιμα, είναι στη διαθέση του κάθε ενδιαφερομένου. Η κοινωνία των πολιτών επίσης με τις οργανώσεις της πρέπει να συμμετέχει στις διαβουλεύσεις και να συμμετέχει με τον τρόπο αυτό στις στρατηγικές επιλογές. Επίσης, λέω ότι θα πρέπει να εξετάζουμε εάν οι επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο μείγμα είναι, έχουν δράση ικανοποιητική ως προς τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Η κυρία Ζόλη φαντάζομαι θα χάρει με αυτό. Θα ελέγχεται δηλαδή εάν πληρούν και τις φορολογικές υποχρεώσεις τους ώστε να μην λησμονούμε και όλη τη συζήτηση για την φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Έχω την αίσθηση ότι η Επιτροπή και οι εδώ παρόντες θα τίνουν ευηκονούς στα όσα είπα γιατί είμαι διτεθμένος να παρακολουθήσω αυτή την υπόθεση και να δω αν υπάρχουν νέα στοιχεία. Δεν ξέρω εάν Κάποιο εκπροσωπεί εδώ την Επιτροπή και θέλει ενδεχομένω να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενημερωτική έκθεσή σας. Ευχαριστώ τον Στέις για την ενημέρωση και τη σημαντική αυτή συνάντηση στην οποία έλαβε μέρος και παρουσίασε συνοπτικά όλες τις αρχές, αρχές δράσης που έχουμε ένας μόνο έχει στήσει το λόγο, ο κύριος Μπέρμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπάρτ, ευχαριστώ πολύ. Και για την επισκόπηση και για το, για το υπόμνημα. Μια ερώτηση μόνο. Χαίρομαι ιδιαίτερος που συζητούμε που το μείγμα αυτό γίνεται τρόπος χρηματοδότηση το 2008 και μου κάνει εντύπωση που χρειάστηκε να περάσει τους χρόνους για να βρεθούν νέα μέσα. Πιέζαμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για νέους, νέες λύσεις. Ε, τελικά τα καταφέραμε. Αλλά κάτι που δεν βλέπω εδώ στο υπόμνημά σου. και είναι το εξής. Το μείγμα δανείων, χορηγιών, επιδοτήσεων θα έχει σημαντική ε, μόχλευση ως προς το κοινό, σημαντική λειτουργία μόχλευσης. Και αυτό για να μην δοθούν ε, άλοφοι στην έλλειπη χρηματοδότηση της ε, ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πάρτεβιτεν, δύο ονόματα ακριβώς ίδια για την ίδια συνέντευξη. Παρακαλώ από την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα... Θα μπορούσα να μιλήσω Ολλανδικά, αλλά θα προτιμήσω τα Αγγλικά. Ε, μια φορά μπορούν και οι Ολλανδοί διερμηνείς να ξεκουραστούν, ε. Όχι, όχι, θα τα πω στα Αγγλικά τελικά. Για τις παρατηρήσεις του κύριου Στάς. Αποτελούν μια καλή καταγραφή της συζήτησης και πρέπει να δούμε ότι το blending platform αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αξιοποιείται, λειτουργεί καλά και μπορούμε και μέσω πρόθεσμα να το εξετάσουμε την ε, Παρασκευή. Συζητήσαμε ένα πρώτο, μία πρώτη αρχική ε, έκθεση και περιμένουμε σε αρχές του 2014 μια πιο διεξοδική περιγραφή με τα όσα θα έχουν προκύψει από τις τεχνικές συζητήσεις και από την ομάδα πολιτικής στο Policy Group. Το Κοινοβούλιο ως παρατηρητής στο Policy Group είναι βεβαίως ευπρόσδεκτο πολλά μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Γραμματείας της έχουν λάβει μέρος και στις τεχνικές ομάδες. Πολλές από τις παρατηρήσεις λοιπόν που επισημάνθηκαν από τον κύριο Στάς χρειάζονται περαιτέρω συζήτηση και μπορούν στις τεχνικές αυτές ομάδες να αναπτυχθούν και μέσα από τις διμερείς επαφές με το Κοινοβούλιο αλλά και στο πλαίσιο αυτής της ομάδας για την πολιτική policy group. Ίσως ήταν υπερβολικό να επισελθώ σε κάθε λεπτομέρεια, αλλά η συμμετοχή των αντιπροσωπιών και της κοινωνίας των πολιτών είναι ως εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αντιπροσωπίες τη συμμετέχει ήδη στα διάφορα έργα και απαιτούμε τα ιδρύματα να προβαίνουν σε τακτικές διαβουλεύσεις, ε, ώστε να τον πιο νωρίς κατά την προτιμωσία ενός ε, έργου με τις αντιπροσωπείες. Ενισχύεται λοιπόν περισσότερο ο ρόλος των αντιπροσωπιών, στόχος κοινό και για την Επιτροπή και για το Κοινοβούλιο και επίσης ε, προκαταβολικά των έργων, ο εντοπισμός δηλαδή των στόχων θα πρέπει και αυτός να γίνεται με βάση τη συνεργασία με τις αντιπροσωπείες. Με τη συμμετοχή αυτών των αντιπροσωπείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω και την ε, δέσμευση της ε, κοινωνίας των πολιτών, της εντόπιας κοινωνίας των πολιτών, ε, αλλά και για το blending και για την πλατφόρμα αυτή τον Απρίλιο. Θέλουμε να συνεχίσουμε τις ανταλλαγές με την κοινωνία των πολιτών για το θέμα του, της στόχιας και την ιδιαίτερη έμφαση που θα δοθεί σε αυτή μας από, το τα blending facilities. Υπάρχουν διάφορες πτυχές εν προκειμένου και κάποιες από τις παρατηρήσεις την ε, εξάντια και εξπόστα αξιολόγηση της φτώχειας, θα πρέπει να δούμε τι είδους συνέπειες μπορεί να έχει, τι μπορεί να προσφέρει, πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί στην πράξη. Και επιπλέον θέλουμε με τα blending facilities πέραν των υφισταμένων τομέων να αναπτύξουμε περαιτέρω και να συνεργαστούμε σε θέματα υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πράγμα το οποίο σφαλώς έχει σημασία για την δημιουργία θεσμοκρασία, τον περιορισμό της φτώχειας, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα στους ε, κοινωνικούς τομείς, όπου είναι αυτό εφικτό βέβαια, και στη γεωργία. Σε αυτά θα περιοριστώ προς το παρόν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ειδικέ ερωτήσεις. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ καθώς ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση, νομίζω ότι πολύ σωστά είπε ο κύριος Μπέρμαν ότι δεν θα πρέπει να καταστεί το mixing αυτό άλοθη για περικοπή ε, κονδυλίων, περιορισμό της αναπτυξιακής βοήθειας. Αυτό μου θυμίζει, για να κλείσουμε με ένα χαριαντισμό, κάποιος είχε πει ότι ο πολιτισμός είναι όπως ε, η μαρμελάδα. Όσο πιο λίγη έχουμε, τόσο περισσότερο την απλώνουμε. Αυτό λοιπόν για να κλείσουμε ένα αστιάκι. Κύριε Στάς, για τα συμπεράσματα. Πρόεδρε. Ναι. Ήθελα να πω ότι βεβαίως αυτό το υπόμνημα είναι ενημερωτικό, έχει ενημερωτικό χαρακτήρα κατά τη συζήτηση, όμως τώρα η ομάδα, η τεχνική ομάδα υπαριθμών 2 κατέθεσε τα επιτεύγματα σε σχέση με αποτελέσματα και μιλήσαμε πολύ για ε, τον τρόπο μέτρησης και αντιλαμβάνομαι βεβαίω το ερώτηση γιατί από την Ολλανδική κυβέρνηση ιδιαίτερα οι εκπρόσωποι έδωσαν, ε, έδειξαν ευαισθησία στα θέματα αυτά. Η κατάσταση κατά χώρες και οι προσπάθειες για περιορισμό της αναπτυξιακής βοήθειας από πλευράς Ολλανδικής κυβέρνησης είχαν σαν αποτέλεσμα από ό,τι κατάλαβα εγώ να προσπαθήσουν οι κάτω χώρες να συγκαλύψουν περισσότερο αυτές τις τάσεις μιλώντας δηλαδή περισσότερο για μείγμα και σας το λέω μια ο Ολλανδούς εσείς κυρία Μπέρμαν δεν έχω τώρα τα, τις σημειώσεις μαζί αλλά την συμπληρωματικότητα την, ε, έθεκ, την έθεξα τη Και πάντως είναι ένα θέμα που πρέπει πολύ προσεκτικά να παρακολουθούμε. Καλώς λέει η Πρόεδρο, στο σημείο 10 τώρα της ημερήσιας διάταξης, εντολή για τριμέρη διάλογο. Η απουσία τελική συμφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για το Πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο έχουμε καθυστερήσει στα πλαίσια της διαδικασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει παρουσιάσει ακόμα σχέδιο προϋπολογισμού. Είπε ότι την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, θα παρουσιάσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που είναι πάρα πολύ κοντά στο σχέδιο θα έλεγε κανείς. Οι συντονιστές της Επιτροπής Προϋπολογισμών αποφάσισαν ότι την 1η Ιουλίου θα υιοθετήσουν ένα σχέδιο εντολής για τον τριμερή διάλογο και η εντολή αυτή θα επιβεβαιωθεί με ένα ναι ή όχι στη συνεδρίασή της της 11ης Ιουλίου. Η κανονική διαδικασία με μια έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και γνωμοδοτήσεις των άλλων επιτροπών δεν ισχύει πλέον εφέτος. Η συνεισφορά της Επιτροπής μας μπορεί να πάρει τη μορφή, πρέπει να πάρει τη μορφή μιας επιστολής στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, στην οποία εξηγούμε τις προτεραιότητές μας. Η συγητής μας είναι ο κύριος Κορτές Λάστρα. Προετοίμασε ένα σχέδιο το οποίο έχουμε ήδη λάβει. Θα προχωρήσουμε σε μια συζήτηση πάνω σε αυτό το σχέδιο επιστολής. Δυστυχώς ο κύριος Κόρτε Λάστρα δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα. Ζήτησε λοιπόν από τον κύριο Μπέρμαν να τον εκπροσωπήσει. Κύριε Μπέρμαν έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα διαβάσω τα, τις σημειώσεις μου στην αγγλική γλώσσα. Αυτές είναι, θα έλεγα, οι σημειώσεις που μου έδωσε ο Ρικάρντο Κόρτες Λάστρα. Εγώ θα συμπληρώσω αυτά που είπε η Πρόεδρος, η πρόταση για την διαδικασία και κάποια σύντομα σχόλια για το περιεχόμενο της πρότασης επιστολής προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών που λάβατε σήμερα το πρωί. Για τη διαδικασία πρώτα. Θα πρέπει, ε, όπως και η Επιτροπή Προϋπολογισμών φέτος, να αυτοσχεδιάσουμε, γιατί δεν υπήρξε ουσιαστικά προσχέδιο. Η συνάντησή μας είναι η τελευταία, πριν χρειαστεί να στείλουμε την επιστολή μας στην Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών. Δεν ξέρουμε ακόμα τι προτείνει ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εισηγητής μας θεωρεί ότι η συνεισφορά μας στον προϋπολογισμό θα είναι αποτελεσματική αν περιλαμβάνει κάποια σχόλια της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα κατατεθεί μεθαύριο ημέρα Δετάρτη. Συζητώντας την πρόταση αυτή με το προσωπικό της ομάδας και της Επιτροπής μας το ταχύτερο δυνατόν, και δίνοντας την δυνατότητα στη γραμματεία μας να διατυπώσει την επιστολή, θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς το ταχύτερο δυνατόν στις εργασίες της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Λοιπόν, αυτό προτείνει ο Λάστρα. Περιμένουμε δύο μέρες, παίρνουμε την πρόταση της Επιτροπής και τη σχολιάζουμε. Τώρα, στα πλαίσια του δημοσιονομικού τριμερούς διαλόγου. Ε, το μέγεθος των πιστώσεων αν θέλετε είναι αυτό που έχει σημασία. Εμείς θα πρέπει να υπερασπιστούμε τα επίπεδα χρηματοδότησης για την αναπτυξιακή βοήθεια και την ανθρωπιστική βοήθεια. Και αυτό θα πρέπει να είναι το κεντρικό χαρακτηριστικό της επιστολή μας στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Οι συζητήσεις σήμερα γίνονται για περικοπές, για περιορισμούς, για παγώματα πληρωμών αλλά δεν υπάρχει δικαιολογία να εξοικονομήσουμε, για να εξοικονομήσουμε χρήματα στις πλάτες των φτωχότερων και των πλέον αδύνατων. Έχουμε πάντα τους ιδίους στόχους που είναι κυρίως η ε, συρρήκνωση της φτώχειας, γιατί το μέλλον των φτωχών είναι και οι δικές μας αγορές. Δεν πρέπει λοιπόν να αυτοπυροβοληθούμε. Πρέπει να μην ξεχνάμε επίσης ε, και ότι χρειάζονται χρήματα και για κλιματολογικές παρεμβάσεις, για μετρίαση των κλιματολογικών συνεπειών, χρήματα τα οποία θα πρέπει να προέλθουν εκτός του προϋπολογισμού, αλλά να ενταχθούν βέβαια ε, στο σύνολο των πολιτικών μας. η δυνατότητα ανάμιξης δανείων, επιδοτήσεων κτλ. είναι κάτι το οποίο απορρίπτουμε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφέρθηκα άλλωστε σε αυτό στη συζήτηση που είχαμε πριν 10 λεπτά. Μπορούμε εμείς ε, ε, να απελευθερώσουμε κάποια χρήματα υποτίθεται από τις χώρες μέσου επίπεδου. Παρ' όλα αυτά αυτό δεν είναι αλήθεια όπως σας είπα γιατί η φτώχεια σε αυτές τις χώρες είναι πάρα πολύ μεγάλη και πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και να μην θυσιάσουμε τις μέχρι τώρα προσπάθειες. Εμείς θα πρέπει βέβαια τις προτάσεις μας να τις κάνουμε παρότι η κριτική είναι ισχυρή εις βάρος τους, υπάρχει υποστήριξη όμως από την κοινή γνώμη. Όταν έχουμε την πρόταση της Επιτροπής λοιπόν για το 2014 θα μπορέσουμε να στείλουμε ένα ισχυρό θα έλεγα μήνυμα προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών προς την κατεύθυνση που προανέφερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέρμαν. Θα ήθελα κάποιος να πάρει το λόγο για τον προϋπολογισμό του 14. Ελπίζω όχι, λέει ο κύριος Μπέρμαν. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Ευχαριστώ. Είπαμε ήδη ότι το βασικό ζήτημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταθέσει ε, πριν από την 1η Ιουλίου μια πρόταση και την Τετάρτη θα καταθέσει την πρόταση Επίτροπός μας. Δεν έχουμε επιπρόσθετα σχόλια προς το παρόν. Euh, Κύριε Μπέρμαν, συμπεράσματα. Ε, <laughs> υπάρχει ελπίδα. Μάλιστα. Το καταγράφουμε, λέει η Πρόεδρος, ότι υπάρχει ελπίδα ακόμη, ότι δεν θα περικοπεί ο προϋπολογισμός μας και οι πιστώσεις, κυρίως για την κατεπίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα αποθεματικά λόγω της διεθνούς κατάστασης ε, που είναι τέτοια ώστε δεν μπορούμε να προβλέψουμε μείωση των αναγκών. Ευχαριστώ σε όλους. Θα περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Πρέπει να βγάλετε τις κάρτες σας για να κάνουμε μια δοκιμή. On a le euh,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

Εξακολουθεί να λείπει μία ψήφος. Tu crois. Καλά πέρας ψηφοφορίες για να δούμε και ας περάσουμε στην κανονική ψηφοφορία. Τι ψηφίζουμε πρώτα, το πρωτόκολλο Κυριμπάτη Ευρωπαϊκή Ένωση Είναι έκθεση του κυρίου Νόισερ. Ψηφίζουμε την πρώτη τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τροπημένο κειμένο υπέρ. Κατά. σε εγκρίνεται. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. 16 με την κυρία το Ιεριπέρ. 4 κατά. Καλά, θα μας το λέτε προφορικά. Κατά είμαι. Ωραία, πέντε ψήφι κατά. Ευχαριστώ. Peut-être. Pouvez-vous mettre Oui, mettez-vous à un autre endroit. Alors, donc, nous allons maintenant voter le rapport de M. Kaminski. Alors, amendement... Θα ψηφίσουμε de εκθέση Kaminski. τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία. Προφορική. Τρία. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αμάνμα. Τέταρτη τροπολογία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 5. Άρχεται. και κλώ. Πέρας. Απορρίπτεται με ισοψηφία. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία για 7. Ε, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά αποχές κρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές κρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά Άποχες εγκρίνεται. Μέχρι την 18, 16, 17 και 18 μπορούμε... Α, δεν μπορούμε. 16 λοιπόν υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. 20. δεύτερο τμήμα. Επαλήθευση ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 21. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι. Καλά, συγγνώμη, δεν, δεν είδα. 21, το δεύτερο τμήμα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας.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 Συγχαρητήρια κύριε Τόμας Καμίνσκι. Alors, nous allons vérifier, nous allons maintenant voter l'avis. Θα ψηφίσουμε τώρα την γνωμοδότηση του κυρίου Κασμάρα και ντροπή τη οδηγία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ποιότητα των καυσίμων και την ε, οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Tu me dis quand ça sera le moment. Je comprends pas. Bon. Donc, euh, amendement. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Επαληθεύουμε. Άρχεται η σωφορία πέρασε. Απερίφθη. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται συμβαστική πρώτη υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 14 σε τμήματα πρώτο υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απερίφθη. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. Δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 18 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Υπέρ τρα κατά αποχές εγκρίνεται όχι επαληθεύουμε ηλεκτρονικά πέρας απερίφθη Στο συγγνώμη 23 τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Είκοσι τέσσερα υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κατά αποχές εγκρίνεται τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τριάντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δύο υπέρ κατά αποχές απερίφθη. πέντε υπέρ κατά άποχες απερίφθη. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 σε τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές απερίφθεια Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά αποχές επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Μα λείπει μία ψήφος. Πέρας ψηφοφορίας. Απερίφθη. 41 υπέρ. Α, σε δύο τμήματα η 41. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. 42 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 43 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 44 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Πέρας. Απερίφθη. Σαραντοχτώ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 48 ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απερίφθη. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε ηλεκτρονικά την 53. Πέρας. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Στο σύνολο. Της γνωματότητας όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχουμε τρει... Donc, ça donne... Ηλεκτρονικά λοιπόν 20 υπέρ, 1 κατά, 3 αποχές. Και συγχαρητήρια στον κύριο Κάσμαρεκ. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, il n'y a pas de questions d'hiver. La date de notre prochaine réunion est le mardi 9 juillet. Προσεχή σε 9 Ιουλίου, Τρίτη, από τις 9 μέχρι το 10.30 και από τις 3 μέχρι τις 6.30. Εμείς δε, θα ασχοληθούμε με το DCI με την ε, κυρισμένη των θηρών συνεδρίαση.